Good morning everybody. Καλημέρα σας σε όλους αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι σας φυσικά. Full house this morning. Είμαστε πλήρης στην αίθουσα και έχουμε το όλο τον κόσμο για τις πολύ σημαντικές ψηφοφορίες που θα λάβουμε χώρα. Έχετε τις ε, κάρτες ψηφοφορία σας. Θα τις χρειαστείτε. Σημείο 7 της ημέρησης διάταξης. Τροποποίηση του κανονισμού 2002 σε σχέση με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Ο Μπαρτ Στάς είναι ο εισηγητή. Περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 26. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 7 εκπίπτει. 27 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 88 με προφορική τροποποίηση και χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά άποχες δεκτή. Εκπίπτει ψηφοφορία κατά κομμάτια. 29 Φερέρα ψήφι ψηφίπερ Για την 29 κατά. Άποχες δεκτή. 8 ψήφι ΠΕΡ, Εκπίπτει. Μάλιστα. 9 υπέρ. Για την 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 έχει αποσυρθεί. 30 ψήφι Κατά. Αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή η 12 έχει αποσυρθεί 32 με προφορική τροποποίηση ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ Κατά. Αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές δεκτή. 14 εκπίπτει. 35 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή αιτιολογικές σκέψεις 15 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή η 1 έχει αποσυρθεί. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές δεκτή. 20 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές γιατί δύο ναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Απόχες δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Απόχες δεκτή. 5 ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες εντάξει δεκτή. 6 έχει αποσυρθεί. 25 ψήφι υπέρ Κατά. Αποχές δεκτή. 23. Υπέρ. Με προφορική τροποποίηση και χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ξεκινάμε με το πρώτο μέρος. Δεν, όχι, όχι σε χωριστά μέρη. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελεκτρονική τελική ψηφοφορία, παρακαλώ ψηφίζουμε. ένας ε, από το ΕΛΚ ε, επιπλέον που ψηφίζει παραπάνω από αυτού που επιτρέπονται και ένας ε, μη εγγεγραμμένο. Α, ακόμα ένας μη εγγεγραμμένο. Και από το ΕΛΚ ακόμα ένας παραπάνω. Θα πρέπει να αποσυρθούν, πρέπει να <laughs> συνηθίσουμε σήμερα. Λοιπόν, ένας μη εγγεγραμμένο να αποχωρήσει και ένας του ΕΛΚ να αποχωρήσει. Να, ένα επιμένει όμω. Ποιο είναι μη εγγεγραμμένο από εσά, Σε σα. Ακόμα, ακόμα είναι ένας ε, υπεράριθμος. Μπορούν οι μια εγγεγραμμένοι να συμφωνήσουν ποιο θα πρέπει να αποσυρθεί. Εντάξει. Αλλά τώρα έχουν προσθέσει πράσινοι ένα, ένα κόμμα που ψηφίζει. Λοιπόν, περιμένουμε. Α, ωραία, εντάξει, τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα είμαστε εντάξει. 58 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε ιδιαίτερα τον κύριο Μπαρτ Στάς. Σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. 8. Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Η συζητήτρια είναι η Ρενάτε Ζώμα. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ. Κατά Απόχε. Και αυτή δεκτή. Συ... Παγιοποιημένη τροπολογία υπεριθμών 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την παγιοποιημένη 4. Το ΕΛΚ έχει τρεις υπεράριθμους, λέει ο πρόεδρος. Και ο κύριος Χάρτουγκ περισσεύει στους ε, μη εγγεγραμμένου. Πρέπει να βγάλει την κάρτα του. Το κόμμα ένα παραπάνω, δύο παραπάνω. Η φιλελεύθερη ένα παραπάνω. Το ΕΛΚΑ ένα παραπάνω. Η φιλελεύθερη ένα παραπάνω. Ε, εξακολουθείτε. Είναι εντυπωσιακή η, η προσήλωση στην ψηφοφορία, αλλά περισσεύει κάποιο Φιλελεύθερη πάλι περισσεύει ένας. Ο Νιούτον Ντάν αποσύρθηκε, το ΕΛΚ ακόμα έχει ένα παραπάνω. Εντάξει. Κάποιος συντονιστής θα πρέπει να επιβάλλει την τάξη στην ομάδα του. Εξακολουθείτε να είσαστε πάνω από το κανονικό όριο. Λοιπόν, εντάξει, πέρας, πέρας 36 υπέρ, 23 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται η παγιοποιημένη 4. Οπότε εκπίπτει η παγιοποιημένη 5. Πάμε στην παγιοποιημένη 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Έλεγχο, έλεγχο βεβαίω Για την 6. Ε, Σοσιαλιστές και ΕΡΚ έχουν ένα παραπάνω. Το ΕΛΚ έχει ακόμα ένα παραπάνω. Ακόμα. Ο Πέτερ Λίζε φταίει για όλα αυτά. Μήπως ε, μπορείτε να πείτε ποιος από εσά δεν θα ψηφίσετε. Είσαστε ακόμα παραπάνω. Είσαστε... Λοιπόν, εντάξει. Τέλος ψηφορία. 29 υπέρ, 32 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται η παγιοποιημένη έξι. Παγιοποιημένη 7, ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. Συνεχίζουμε λοιπόν. 137. Με χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος βεβαίως. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, ναι, σαφώς απορρίπτεται. Όταν βλέπω έτσι την πλειοψηφία είναι σαφές ότι είναι έτσι. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Ψήφι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά. Αποχές δεκτό. Είκοσι με χωριστή πάλι ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 138 με την ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το πρώτο τμήμα τη 138. Το ΕΛΚ έχει ένα με υπερβάλλοντα ζήλο πάλι. Εντάξει τώρα, πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. κατά αποχές δεκτή. 139 και 140 είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 1.41 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά <clears throat> αποχές δεκτή. 142, 143, 144 που είναι ταυτόσιμες ψηφίτε κατά αποχές δεκτή. Δεκτές. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 145 υπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος, βεβαίως, με 145. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 29 σε δύο τμήματα. <clears throat> Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 30α και 147 ταυτίζονται ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτές. 300 πόσο λέει ο πρόεδρος 30 β <laughs> συγγνώμη 30 β ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος στην 30 β ηλεκτρονικός Οι σοσιαλιστέ έχουν ένα που περισσεύει. Εντάξει τώρα. Πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται. 31. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 149 υπέρ. 32 θέλετε έλεγχο. Εντάξει, 32 έλεγχος. Πέρας. Δεκτή 32. 149 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Σαφές για μένα, αλλά μα θέλετε κάνουμε έλεγχο για την 152. Ε, Σλούτερ Ριβάζη. Πέρας προφορίας. Δεκτή. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 151 και 153 είναι ταυτόσιμες υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Απορριπτονται. Συνεχίζουμε. «33 ψήφι υπέρ». «35 μάλλον υπέρ». «Κατά». «Αποχές απορρίπτεται». «37 υπέρ». «Κατά» αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> Έλεγχος. Για την 155. Πέρας ψηφοφορίας. Σαφώς εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για 158 απορρίφθηκε, εντάξει. 39. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για τις 40. Πέρα στις πληροφορίες Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 141 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λοιπόν, με την 187 πάμε τώρα. Καρτή Λιωτάτ. Ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 συγγήτριες. Πέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 189 και 190 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτή. 49 εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτει. Έλεγχος για την 49. Ε, Πέρας. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Πέρας. Δεκτή. 139. Έχουμε καταρχήν την προφορική τροποποίηση. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροποποίησης. Κατά. Αποχές δεκτή. Η τροπολογία πως έχει τροποποιηθεί. 193 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 194 και 192 είναι ταυτόσιμες αλλά εκπίπτουν μετά την έγκριση 193, σωστό. 51α χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Εκπίπτει. Ευχαριστώ κύριε Συγήτρια. Το δεύτερο τμήμα και το πρώτο τμήμα λύση η Όχι, όχι, μόνο το δεύτερο τμήμα εκπίπτει, λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα τη 51α. Πρώτο τμήμα, λοιπόν, ψήφι υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές δεκτό. 194β ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Έλεγχος, έλεγχος για την 194 β. Πέρας της Στο τσακ εγκρίνεται. 195 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έλεγχος στην 195. Πέρας προφορίες. Εγκρίνεται. Σαφώς. Εκατόν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ...205 της εισηγήτριας, ψήφι υπέρ. Κατά, άποχες, δεκτή. 209 υπέρ. Κατά, άποχες, δεκτή. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πηδάμε κάτι σελίδες. για μένα είναι η σελίδα 13. Είναι η τροπολογία 56. Τη βρήκατε, τη βρήκατε, ψήφι υπέρ. Όχι ακόμα. Άρθρο, άρθρο 26 παράγραφος 1, τροπολογία 56, εκεί είμαστε, σελίδα 13 στο αγγλικό κείμενο, ψήφι υπέρ, κατά, κυρία Βίλματ. Πηδήσαμε ορισμένε ε, τροπολογίε, αλλά οι 2.14, 2.17 και 2.23 πρέπει να εκπέσουν εάν περάσει παγιοποιημένη 4 είπατε, αλλά είναι ειδικέ ψηφοφορίε. Δεν νομίζω ότι καλύπτονται από την παγιοποιημένη τροπολογία, ούτε είτε ο σκοπό αυτή τη τροπολογία να τι καλύψει. Εγώ θα πρότεινα το εξή. Νομίζω ότι η εισηγήτρια διαφωνεί. Θα πρέπει να ψηφίσει η Επιτροπή μας κατά πόσο πράγματι καλύπτονται οι τροπολογίες αυτές ή όχι. Λοιπόν, πρέπει να διαβάσουμε τώρα να δούμε τι λένε οι τροπολογίες. Μπορεί να μας αναφέρει πάλι τις τροπολογίες η κυρία Βίλμοντ. Πεςτε μας ποιες είναι οι τροπολογίες που νομίζετε ότι πρέπει να ψηφιστούν η τροπολογία 21 στο άρθρο 25 παράγραφος 2, η 200, συγγνώμη, η 214 στο άρθρο 25 παράγραφος 4, η τροπολογία 214. Δεν καλύπτεται κατά την άποψή μου. Καθώς και 217 και 223 λέει η κυρία Βίρμοντ Λοιπόν, επειδή είναι ταυτόσιμες, τις διαβάζω. Το κείμενο λέει, όταν υπάρχουν λόγοι που θα καθιστούσαν μη πρακτικό να υπάρχει ετικετοθεσία για τη χώρα προέλευσης για το κρέας και τα πολερικά σε ε, επεξεργασμένα τρόφιμα θα μπορούσε να γίνεται η εξής δήλωση ε, μέσα σε, σε παρένθεση μη γνωστής προέλευσης. Αυτό λένε οι τρεις τροπολογίες για τις οποίες να, θέλει η κυρία να ψηφίσουμε η συγγήτρια και μετά θα πρέπει να ψηφίσουμε. Παρακαλώ κυρία Ζώμερ. Όσο και να το <clears throat> έτσι θα περάσουμε μέρες να ελέγχουμε τι καλύπτουν ή δεν καλύπτουν οι παγιοποιημένες τροπολογίες, λέει η κυρία Ζώμερ. Οι τροπολογίες αυτές δεν πρέπει να προσθεθούν επιπλέον, γιατί πράγματι εκπίπτουν μετά από την έγκριση της παγιοποιημένης τροπολογίας υπαριθμών 4. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εντάξει, λέει ο πρόεδρο, ας ψηφίσουμε. ποιο θέλει να ψηφίσουμε αυτές τις τρει επιπλέον τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. Πάλι πρέπει να κάνουμε και έλεγχο λοιπόν για αυτή τη διαδικαστική πρόταση. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ ή κατά θα πρέπει να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Πέρας. Λοιπόν, απορρίπτεται η διαδικαστική αυτή πρόταση. Δεν θα ψηφίσουμε αυτέ τι τροπολογίε. Είμαστε λοιπόν στην 56. Ψήφι Κατά. Αποχές δεκτή. 269. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.70 και 2.74 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή, δεκτές. Έλεγχος βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. με μία ψήφο διαφορά. Απορρίπτεται, βλέπω δεν ψηφίσατε όλοι βέβαια αυτή την τροπολογία, αλλά απερίφθη. Τι να κάνουμε. 276 2.71 από κοινού ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας πληροφορίες. Ενέκρινται. Μάλιστα. Οπότε προχωράμε στην 57β. Ψήφι 57β. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 57β. Πέραση της ψηφοφορίας. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα που περισσεύει. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτή. 2.77, 2.78 είναι ταυτόσιμες και 279 επίσης ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομίζω ότι είναι σαφές, δεν χρειάζεται έλεγχο. Κύριε Χάρτον, πρέπει να βγάλετε την κάρτα σα. για τον ηλεκτρονικό έλεγχο, πέρα του ελέγχου, δεκτή πράγματι. 57α και 280 που ταυτίζονται, ψηφιπέρ. Κατά. Δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ λίγοι ο τα χέρια. Πάλι ψηλά τα χέρια. 57α και 280. Ψήφι υπέρ. Τώρα ναι φαίνεται. Κατά. Αποχές δεκτή. 281 καθώς και 282 που ταυτίζονται. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεκτές. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δύο <clears throat> υπέρ, κατά 285 λοιπόν. Λοιπόν, αν θέλετε κάνουμε έλεγχο. Νομίζω ότι είναι σαφές το αποτέλεσμα για την 59. Κάνουμε έλεγχο για την 59 πρώτα. «59, εντάξει, έλεγχος». Τέλος. Κάτι, κάτι δεν πήγε καλά. Η κυρία Ζόμερ ζήτησε έλεγχο για την 59, που είναι τροπολογία διαγραφής του άρθρου 29. Άλλη μια φορά από την αρχή. Τροπολογία 59, άρχεται η ψηφοφορία. 59, όχι τίποτα άλλο. Πέρας. Απορρίπτεται λοιπόν. Τώρα πάμε στην 285. Λιωτάρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 287 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 62, 63, 64 αλλά και 65 unblock, μπλοκ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 2,88 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Πέρας <coughs> ψηφοφορίας. Δεκτή. 289 <coughs> υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορριπτή. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Σε χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος. Λοιπόν, πρώτο μέρος 290 υπέρ, κατά Αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα. Έτσι πρέπει να ψηφίσουμε όλες σε κάθε σημείο ξεχωριστά διότι απορρίφθηκε μια παγιοποιημένη η 291 υπέρ 291 ναι έχει το λόγο όχι όχι πέστε μας Νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος στον κατάλογο αυτό ψηφοφορίας. Εδώ μιλάμε για τη 291, η οποία έχει καταπέσει όμως από τη στιγμή που η 6 έχει υιοθετηθεί. Η 7 έχει υιοθετηθεί και αυτό ήταν ε, άλλη προϋπόθεση για να καταπέσει αυτή εδώ. Άρα λοιπόν η 291 καταπίπτει από τη στιγμή που η 7 έχει υιοθετηθεί. Αυτά. Όχι, δεν, η γνώμη μας δεν είναι η ίδια. Θα ψηφίσουμε εδώ. Ψηφίζουμε για αυτήν. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε. Ένα το ΕΛΚ επιπλέον παραπάνω, εντάξει αποσύρθηκε, τελειώσαμε. Η πλειοψηφία δεν θέλει να ψηφίσουμε για την 291. Για να δούμε. Ε, διαδικαστικό, Σλίτερ. Ακούστε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να ψηφίσουμε. Υπάρχουν διαφορετικά άρθρα. Η συμβεβαστική 7 αφορούσε το 33. 1 και 2 όμως. Η παρούσα αφορά το 33. 3 Είναι διαφορετικό άρθρο. Χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, Νομίζω όμως ότι ψηφίσαμε, η πλειοψηφία είναι κατά. Πηγαίνουμε στη 292 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 293 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. ένας πάλι παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 297 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 297 ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα 294, 295, 298, 300 ταυτόσημες, 300 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Απορρίπτεται. 301 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 299 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε αν θέλετε ηλεκτρονικά. 71 λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Υιοθετείται. Εγκρίνεται λοιπόν. 71. Προχωράμε. 73. 33. 4. 73 λοιπόν. Υπέρ. Υπέρ της 73. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 312. Προφορική. Υπέρ. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει, απορρίπτεται, απορρίφθηκε μάλλον. Ψηφίζουμε στο αρχικό κείμενο, το οποίο όμως αποσύρθηκε. 76α προφορική, υπέρ της 76α, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 313, καταπίπτει αυτή. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρακόσια δεκαέξι. Υπέρ της 316. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 317 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. 76 β. Μάλλον ε, γ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 76 σ. 76 γ λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 318 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε όμως. Ελέγχουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 77. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 320 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 321 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 322 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 323 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 324 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 325 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 80, 81. Ψηφίζουμε. πέρασε Απορρίπτεται. Απορρίπτεται η 81. 326 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι 326 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ένας από τους σοσιαλιστές είναι παραπάνω πέρας απορρίπτεται 82 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 327 καταπίπτει. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 83 παρακαλώ. Ε, κα, όλο και κάποιος μας λείπει τώρα. Για να δούμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 330 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 329 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 331 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 332 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 333 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 334 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 335 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 336 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 337 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 338 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 341 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 342 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 343 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 344 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 345 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 346 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 347 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 348 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 349 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 350 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 350. Για την 350 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 351 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 353-359 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Σε δύο χωριστά μέρη 355, η πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ναι. Σωστά. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 356 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 352 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 357 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 358 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 360 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. 96 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Σαφώς εγκρίνεται. Η επόμενη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 363. 362-64 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 366 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 366. Πέρας. Εγκρίνεται σαφώς. Εγκρίνεται. Τώρα να συνεχίσουμε 373, 370, 371 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας, εγκρίνονται. 381 προφορική τροπολογία υπέρ παρακαλώ αυτής της προφορικής τροπολογίας 381 κατά να ελέξουμε ηλεκτρονικά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την, ηλεκτρική, για την ε, προφορική τροπολογία 381 Πέρασε. Εγκρίνεται. «382» υπέρ της 382 κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 383 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέξουμε. Να ελέγξουμε για την 383. Πέρας εγκρίνεται. ...384 και 85 και 365 υπέρ αυτών των τριών κατά αποχές εγκρίνονται. 99 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 9. Πέρας. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 387, 388 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. ...386 καταπίπτει, 389 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 390, 391, αυτές οι δύο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται 392, προφορική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 393 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 400. Α, λησμόνισα την 102. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 400 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 401 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δυστυχώς, δυστυχώς λέγω. Κύριε Ντελάγκη, απορρίπτεται. Λοιπόν, 402 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ με την 106 και 107 υπέρ αυτών των τροπολογιών κατά αποχές ε, δεκτές 105 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή αιτιολογικές σκέψεις 1 ψήφι υπέρ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 Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 108. Με χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 109 <clears throat> ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την έξι πέρα της προφορίες. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 110 με χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα. Κατά, αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 9, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Εδώ Υπέρ, κατά, 112 αποχές δεκτή. Οι 10 και 114 που ταυτίζονται υπέρ 10 και 114 κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνονται. 11 υπέρ. Κατά. Άποχες. απορρίβεται 115 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 116 εκπίπτει, 117 υπέρ. κατά άποχες δεκτή 119 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 120 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 122 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124 με χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 128 υπέρ κατά άποχες θα ελέγξουμε την 128 128 έλεγχος Abstimmung beendet. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 10... Η 13. Ψηφίζουμε 13. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά <clears throat> αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές έλεγχος και την 131 Ένας περιπλέον από το ΕΛΚ. Εντάξει τώρα. Πέρα τις προφορίες εγκρίνεται. 131. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 19. Υπέρ κατά άποχες δεκτή. 135 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 136 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Φτάσαμε στην τελική ευθεία, τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο συνολική ψηφοφορία όπως έχει τροποποιηθεί το κείμενο. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας. 57 υπέρ, 4, 4 ψήφοι κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια την κυρία, στην κυρία Ζόμερ για την τόσο σημαντική αυτή η έκθεση. Συγχαρητήρια κυρία Ζόμερ. Ήταν μια μεγάλη μάχη που δώσαμε αλλά έχουμε φτάσει στο τέλος και τώρα η κυρία Βέστρου θέλει να λάβει το λόγο. Eh, θα ήθελα να ζητήσω από τη Γραμματεία και από τον Πρόεδρο να μας πει ποιος κανονισμός εφαρμόζεται όταν ακριβώς αποφασίζουμε για να δούμε ποιες είναι οι τροπολογίες που καταπίπτουν και ποιες όχι. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν υποβάλλει κάποιος μία τροπολογία θέλει να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία του και αν κάποιο μπορεί να πει εντάξει ίσω. Ε, όχι όχι κάποιο ίσω πει δεν την ψηφίζουμε αλλά χωρί να αιτιολογήσει αυτή την απόρριψη τη πληροφορία. ε, δεν ξέρω πρόκειται για μια μέθοδο κάπω παράξενη ειδική. Θα ήθελα λοιπόν ο πρόεδρο μας να συντάξει ένα κώδικα συμπεριφοράς πάνω στο θέμα αυτό για να ξέρουμε τι γίνεται με τι τροπολογίε αυτέ. Γιατί τώρα το να ψηφίσει κανεί αν θα ψηφίσει ή όχι αυτό μου φαίνεται σαν διαδικασία διαδικασία, κάτι που δεν μπορεί να το δεχτούμε, έτσι. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν είναι η συγγήτρια η οποία αποφασίζει, αλλά η... ο κανονισμός του Κοινοβουλίου αποφασίζει για το θέμα αυτό. Και ο κανονισμός του Κοινοβουλίου λέει ότι η απόφαση αυτή είναι στην αρμοδιότητα του Προέδρου ε, της Επιτροπής και σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής. Πάμε τώρα στο ΑΕΠ και επέκεινα είναι η έκθεση της Άννας Ρόσπαχ, παράγραφος 1, τροπολογία έκον 1. Ah also es gibt den Konsens, dass Υπάρχει γενική συνένεση η εισηγήτρια και οι σκιώδεις εισηγητές συμφωνούν να ψηφίσουμε από κοινού τις παραγράφους. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει καμία ε, αντίρρηση, όλες οι παράγραφοι και μετά να ψηφίσουμε μονάχα την τελική ψηφοφορία. Έχετε κάποια αντίρρηση? Ποιοι είναι υπέρ της, ψήφιση υπέρ όλων των παραγράφων που αναφέρονται στο έγγραφο ψηφοφορίας. Κατά. Άποχες. Δεκτές οι παράγραφοι αυτέ. Και ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα. Η κυρία Χάουγκ. Συγγνώμη. Έχουμε ψηφίσει όλες... Έχουμε ψηφίσει ότι θα ψηφίσουμε unblock τις παραγράφους. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε όμως. Και μόνο θα έρθει η τελική ψηφοφορία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να δώσει μια σαφήνεια στην κατάσταση αυτή. Τι ακριβώς ψηφίσουμε unblock. Να μας πει η εισηγήτρια παρακαλώ. Για να είμαστε σύντομοι. Έχουμε από την Οικονομική Επιτροπή, από την Ήτρε και από άλλες επιτροπές έχουμε ψηφίσει τα, τις γνωμοδοτήσεις τους μεταξύ των σκιωδών εισηγητών υπήρξε συμφωνία και είπαμε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Θέλουμε σήμερα απλώς να εκπονήσουμε το έγγραφο βάσης. Και επομένως ζητήσαμε από τους συντάκτες των τροπολογιών να αποσύρουν τις τροπολογίες τους, ώστε σήμερα να καταλήξουμε με ένα ισορροπημένο έγγραφο βάσης. Αυτός είναι ο στόχος. Οπομένω, είπαμε, οι τροπολογίες ΕΚΟΝ, και τα κτλ. να μην ψηφιστούν στη, στην, πρώτη, στην πρώτη ψηφοφορία και να έχουμε ένα κείμενο το οποίο προσωρινά θα είναι το έγγραφο εργασία μας. Εντάξει. Επομένως ψηφίζουμε, όλα αυτά τα οποία είναι σε θεό χρώμα στο φύλλο ψηφοφοριών. Αυτές θα ψηφίσουμε από κοινού, unblock. Και ξαναλέω, ποιοι ψηφίζουν υπέρ των τροπολογιών που είναι σε γκρι χρώμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Α, τώρα κατάλαβα. Αποχές. Ωραία. Πάνε αυτές, φύγανε λοιπόν. Ευχαριστώ Γιούτα. Έχουμε λοιπόν την τελική ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ τη ούτω τροποποιητής ηλεκτρονικά. Παρακαλώ βάλτε τις κάρτες σας. Βγάλτε τις κάρτες σας. Πέρα τη ψηφοφορία. 59 ψήφοι υπέρ, μία ψήφο, κατά, μία αποχή, εγκρίνεται η έκθεση τη κυρία Ρόσπαχ. Συγχαίρω την κυρία Ρόσπαχ για το ΑΕΠ και το επέκεινα του ΑΕΠ. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές, τη γραμματεία, για την έγκριση αυτών των εκθέσεων και περνάμε τώρα. Μάλιστα. Διακόπτει ο πρόεδρος ε, προσωρινά. Έχουμε τώρα ένα σημείο στην ημέρηση διάταξη το οποίο αντιμετωπίσαν χθε οι συντονιστέ και υπήρξε συμφωνία από του σημείου αυτού. 26 Απριλίου είναι τα 25 χρόνια της επαιτίου του ατυχήματος του Τσέρνομπιλ και είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια ερώτηση, προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια και να είναι αποτέλεσμα, αντικείμενο συζήτηση με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Σας έχει διανεμηθεί αυτή η ερώτηση. Έχουν συμφωνήσει αυτοί που υπέβαλαν αυτή την ερώτηση για το κείμενο και θα πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της ερώτησης. Ποιοι είναι υπέρ της υποβολής της προφορικής αυτής τροπολογίας, ποιοι είναι υπέρ του κειμένου αυτού. Κατά αποχές θα ε, υποβληθεί λοιπόν στην Ολομέλεια αυτή η προφορική ερώτηση. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης. Η έκθεση Ορέστη Ρώση. Γνωμοδότηση για την κινητικότητα και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία. Ο εισηγητής, ο κύριος Ρώση, έχει το λόγο. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως και συνάδελφοι, πρόκειται για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση πέρα από πολιτικά θέματα τώρα. Είναι κάτι υπέρ μιας κατηγορίας ε, ατόμων που έχουν προβλήματα και είναι για την απασχόληση και κοινωνική υποθέτηση. είναι η κινητικότητα και η ένταξη αυτών των ατόμων ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020. Άρα λοιπόν αφορά τα επόμενα 20 χρόνια είναι θεμελιώδη σημασία για κάποιον ε, που προχωράει σε αυτού τους κανόνες πάνω σε αυτά τα θέματα, Όπω θέλουμε τα λέμε αυτά τα άτομα με αναπηρίε με προβλήματα κλπ. Ε, πρέπει να έχουν ε, τα ίδια δικαιώματα όπως και οι υπόλοιποι πολίτε. Τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Να ζητήσουμε ακριβώ να καταβάλουν προσπάθειες στα κράτη-μέλη ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητε υπηρεσίε για την διακίνησή του. και να Έχουμε τα ηλεκτρονικές ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και για τις οικογένειες αυτές ε, που προσπαθούν να κρατήσουν μαζί τους αυτά τα άτομα με προβλήματα και να ε, σε οργανισμούς και δημόσιους και ίσως και ιδιωτικούς να παρέμβουμε ώστε να υπάρχουν θέσεις που να αφορούν αποκλειστικά εκείνους που έχουν αυτά τα προβλήματα γιατί έτσι αν ενταχθούν αυτά τα άτομα με προβλήματα, με αναπηρίες σε ένα ενεργό κοινωνικό περιβάλλον, εργασία, ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση, αθλητισμός να μπορούν να κινηθούν με λιγότερες δυσκολίε, σημαίνει αυτός ο κόσμος να έχει τα ελάχιστα απαραίτητα για να ζει καλύτερα να υπενθυμίσουν αδέλφους όλα τα κράτη-μέλη μαζί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν την ε, Σύμβαση των Μενεθνών για τα δικαιώματα αυτών των ατόμων με προβλήματα και αναπηρίες. λοιπόν και εκεί 16 κράτη-μέλη ήδη πριν από λίγα χρόνια υιοθέτησαν αυτή τη σύμβαση και στα υπόλοιπα ε, κράτη προχωράει αυτή η ε, αποδοχή. Και επίση θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλε υγειονομικέ υπηρεσίε για αυτά τα άτομα με αναπηρίε. Γιατί ακόμα και σήμερα από το ένα κάτω στο άλλο υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Θα πρέπει να ε, αποφύγουμε, να δίσουμε τη μάχη μα κατά των προβλημάτων ε, και των ανισορροπιών ε, και να μπορέσουμε να του προσφέρουμε υπηρεσίε κατάλληλε για την ισορροπία του ακριβώ και υπηρεσίε κατάλληλε ώστε να μπορεί κανεί να παρέμβει και μάλιστα από πριν να μπορεί να εκτιμήσει κανεί τι ανάγκε που έχουν αυτά τα άτομα και έτσι να εγγυηθούμε μεγαλύτερη συμμετοχή αυτών των ατόμων με αναπηρίε στα πλαίσια του εργατικού δυναμικού και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τα παροτρύνουμε για να δραστηριοποιηθούν, να συντονιστούν μεταξύ του για καλύτερε πρακτικέ ένταξη και καλύτερε πρακτικέ παρόμοιε για να μην υπάρχουν πια εμπόδια για αυτού. Ένα παρόμοιο άτομο, ας πούμε, που ξεκινάει από το Τωρίνο με ένα τρένο και πάει μέχρι το Μιλάνο θα πρέπει να έχει μόνο δύο τρένα την ημέρα που να έχουν το κατάλληλο σκαλί για να μπορέσουν να ανέβουν. Και ένας πολίτης που φεύγει από την Ιταλία με ένα κατάλληλα τρένο και να φτάσει σε μια άλλη χώρα, έστω και αν υπάρχει αυτό το κατάλληλο σκαλί για να περάσει κλπ. Και, και να υπάρξει πρόβλημα εκεί πέρα, επειδή στην άλλη χώρα δεν υπάρχει κατάλληλη εγκατάσταση. Α, λοιπόν, συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη που είναι κάτι το βασικό. Καταλήγω, ολοκληρώνω εδώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σαν Επιτροπή ε, που ασχολείται και με θέματα υγείας μπορούμε να ενεργήσουμε θετικά υπέρ αυτών που υποφέρουν, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, να τους προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες που και σήμερα ακόμα λείπουν, είτε που υπάρχουν αλλά πάντα με δυσκολίες μεγάλες, μεγάλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Ορέστη. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση που αφορά πολλά εκατομμύρια ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ανάπηρα και αντιμετωπίζουν σε καθημερινό επίπεδο δυσκολίες στη μετακίνησή τους. Και αυτό είναι πολύ καλό αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες μπορεί να πάρει θέση για το θέμα αυτό. Ε, Νέσσερ Τσίλντες έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σκιώδη συγκήτρια για αυτήν την γνωμοδότηση. Θέλω να ευχαριστήσω τον συντάκτη τη γνωμοδότηση. Οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένο ότι μπορούν να ανέβουν σε ένα λεωφορείο ή να πάνε για ψώνια, να επισκεφθούν του φίλου του, να πάνε στο θέατρο, στο σινεμά. Όπως ε, το να ε, ψηφίζει κανείς εκλογές ε, ή να επισκέπτεται το διαδίκτυο. Πάντως υπάρχουν πολλοί συμπολίτε μα που δεν μπορούν, γι' αυτό και αυτή η στρατηγική είναι πάρα πολύ σημαντική για εκατομμύρια συμπολίτε μας. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για κοινωτική δράση στον τομέα αυτό, γι' αυτό θα ήθελα εν συνεχεία να πω ότι Οκτώ βασικούς τομείς δράση έχει εντοπίσει η Κομισιόν. Η δική μας ε, Επιτροπή γνωμοδοτεί, γι' αυτό και εγώ θα μιλήσω για τον τομέα που είμαστε αρμόδιοι, την υγεία. Ξέρουμε ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη ρουτίνας και πρέπει να στηρίξουμε τη λήψη μέτρων ώστε να παρέχονται υπηρεσίες και ευκολίες υγείας χωρίς καμία διακριτική μεταχείριση. Και θέλω να εγκριθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Κάρτα Κινητικότητας που θα είναι αμοιβαία αναγνώριση ε, των εθνικών καρτών αναπηρίας. Και έτσι θα έχουμε αυτή την ε, υποστήριξη για την αρμονισμένη Ευρωπαϊκή Κάρτα. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, συντάξη νομοδότηση που εστιάζει στην υγεία και θα, στη, θα, θα συνεργαστώ μαζί του επόμενε εβδομάδε. κύριο Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και από την ομάδα Άλντε, ακριβώς θα ήθελα να δώσω συγχαρτήρια στον Ορέστη για το πώς συνέταξε την έκθεσή του Νομίζω ταυτόχρονα βέβαια ότι θα δεχτεί και διάφορες αλλαγές τροπολογίες γιατί το θέμα αυτό όπως ακούσαμε έχει σημασία πραγματικά ακριβώς για πολύ κόσμο αλλά κυρίως ε, όχι μόνο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και για όλο εκείνο το χώρο της κοινωνίας που επιδεικνύει μια κάποια ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα ε, του προβλημάτων ε, μετακίνησης ε, και να σας πω κάτι άλλο, ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σε σχέση με προηγούμενες φορές να που προτείνει κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και ενδεικτικό, ότι υπάρχει διάθεση να βοηθήσει και οικονομικά, να υποστηρίξει οικονομικά αυτές τις θετικές ενέργειες, ώστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα να αντιμετωπιστούν ισότιμα τα άτομα αυτά, όχι μόνο όσον αφορά την οργάνωση, αλλά και από κοινωνική πλευράς, ε, για την εκπαίδευση, για την κατάρτιση. Πρόκειται λοιπόν για μέτρο που στο σύνολό του και γενικά είναι υπέρ όλων αυτών που δεν είναι πάντως ίσες δυνατότητες για τους πολίτες που αξίζουν να τους προσέξουμε με τον τρόπο αυτό το θετικό και θα μπορέσουμε να εντάξουμε και νέα στοιχεία έτσι στην έκθεση την οποία και προσεχώς θα υιοθετήσουμε. Να πω μερικά πράγματα προσθετικά. Στο άρθρο 5 ας πούμε της έκθεσης νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ε, για το τι γίνεται με αυτά τα αρνητικά αλλά και προσθέτοντα στοιχεία κατάρτισης εκπαίδευσης για να βοηθήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαμε να υποβάλουμε μια τροπολογία. Επίσης για την κοινωνική προστασία των ατόμων με προβλήματα λείπει κάτι. Χρειάζεται αυτό να το εκφράσουμε ρητά ότι υπάρχει ανάγκη από συστήματος κοινωνικής προστασίας και μείωσης της πτώχειας ας πούμε και κατοικία και διάφορες άλλες υπηρεσίες και επίσης όσον αφορά τις συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Και θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσω επειδή σε αυτά τα προβλήματα υπάρχει και μια διάκριση κοινωνική και επηρεάζει αρνητικά τα άτομα αυτά για την ευμαρία τους. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζονται ενέργειες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να ευαισθητοποιήσουμε κόσμο στις εκστρατείες ακριβώς ευαισθητοποίησης μας απέναντι στους υπόλοιπους πολίτες και να μπορέσουμε να δώσουμε όπως πρέπει τις πληροφορίες που θα βοηθήσουν ε, ε, μέσω κοινωνικών δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συζητούμε ουσιαστικά σήμερα για το κοινωνικό αποκλεισμό όταν μιλάμε για άρση εμποδίων και φραγμών βλέπουμε το πρόβλημα υπό τη σκοπιά, υπό το πρίσμα των φραγμών των εμποδίων. Παραδείγματο χάρη για να μπει κανεί σε ένα τρένο, σε ένα λεωφορείο κτλ. Αλλά αυτά τα εμπόδια δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πρόσβαση. Είτε έχει να κάνει αυτό με τη μειωμένη όραση, είτε με τη μειωμένη κινητικότητα πρέπει να δούμε και τους κοινωνικούς φραγμούς, τα κοινωνικά εμπόδια, παραδείγματος χάρη πρόσβαση στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Υπάρχουν οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, όχι λόγω της ε, ε, οικονομικής τους κατάστασης, αλλά λόγω της δύσκολης πρόσβασης. Επίσης, πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αν υπήρχε δυνατότητα πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασία. δεν θα χρειάζονταν να λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα. Αν είχαμε δηλαδή φροντίσει να υπάρχουν οι όροι και οι συνθήκες ώστε να μην προσφεύγουν στην κοινωνική ε, προστασία, στα κοινωνικά επιδόματα. Και αυτά θα έπρεπε να αποτελούν απλά μια έσχατη λύση. Στόχος μας είναι να διδαχθούμε από την εμπειρία που έχουμε συλλέξει και να στηρίξουμε τελικά τη θέση των ατόμων με αναπηρία. Και αν ε, συνεχίσουμε προς την ε, κατεύθυνση αυτή, νομίζω ότι θα άρουμε όλα αυτά τα εμπόδια, γιατί αυτό είναι εφικτό. Μπορεί να πραγματοποιηθεί. Πρώτη. Να προσθέσω και εγώ κάτι όχι μόνο τα φυσικά εμπόδια αλλά και της επικοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αλλάξει αυτή η τεχνολογία ενημέρωσης και ε, πληροφόρησης για να ξεπεράσουμε και άλλα εμπόδια που είναι ακριβώς επικοινωνίες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά, είναι δυνατό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και σχετικά με κάθε έρευνα και προσπάθεια ξεκινώντας από το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για να ξεπεράσουμε και άλλα επαναλαμβάνω εμπόδια που ισχύουν για τα άτομα με παρόμοια προβλήματα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Επιτροπής από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την εξέταση της ε, ανακοίνωσης για τη στρατηγική δράση ε, στον ε, τομέα της αναπηρίας για την προσεχή δεκαετία. Πολλά σχόλια έχουν επικεντρωθεί σε ειδικέ πτυχές, όλες των οποίων καλύπτονται στη στρατηγική. Η στρατηγική έχει μια ισχυρή εντολή, η οποία σχετίζεται αφενός με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται συνολικά να τηρεί από τον Ιανουάριο ε, του τρέχοντος έτους να τηρεί τις διατάξεις αυτής της σύμβασης. Αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά και την έμπνευσή μας για να διατυπώσουμε αυτή τη στρατηγική με τη λογική της, ε, της συμπερίληψης της διάστασης αυτής σε όλες ε, τις πολιτικές. Θέλουμε να υπάρχει πλήρη συμμετοχή, ένταξη των ατόμων αναπηρία και στην κοινωνία και στην οικονομία. Τώρα, το δεύτερο πλαίσιο, που θέλετε, πολιτικής πρωτοβουλίας αυτής είναι η στρατηγία την Ευρώπη του 2020, όπου τουλάχιστον τρεις από τους βασικούς στόχους για την απασχόληση, την παιδεία και τη μείωση της φτώχειας έχουν πολύ μεγάλη σχέση ε, με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Οι στόχοι αυτοί δεν θα επιτευχθούν εάν δεν υπάρχει πλήρης ένταξη και συμμετοχή αυτού του τμήματος του πληθυσμού και στην οικονομία και στην αγορά εργασίας. Ό,τι αφορά τώρα την προσβασιμότητα, ένα θέμα το οποίο τόνισαν αρκετοί από τους βουλευτές ε, στα σχολιά του σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί πλήρως ότι δεν μιλάμε για φυσικά και περιβαλλοντικά μόνο εμπόδια, υπάρχουν και πολιτιστικά, επικοινωνιακά, κοινωνικά εμπόδια και φραγμοί. Για την αντιμετώπιση αυτών ανακοίνωσε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκπόνηση μιας ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα, η οποία θα ασχολείται ακριβώς με αυτά τα θέματα της πρόσβασης στα αγαθά και στις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Βέβαια, ακόμη είναι πολύ νωρί ε, για να μιλήσουμε για το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά σύντομα θα δρομολογηθεί μια μελέτη για να αξιολογηθούν τα προβλήματα και οι επιπτώσει ε, για τη συλλογή δεδομένων. Και θα ακολουθήσει ευρεία διαβούλευση με ένα ευρύτατο φάσμα εμπλεκομένων, ε, παροχή υπηρεσιών, ε, κλάδος, ε, αρμόδιος και υπόλοιποι, ώστε να έχουμε μια πρόταση να διατυπώσουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή, αν θέλει να μας κάνει και τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ιδιαίτερα ικανοποιημένο είμαι και όλοι οι συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο νομίζω ότι συμβαδίζουν με τους στόχους και βέβαια στο σχόλιο της Επιτροπής ε, αυτό που είπε και αυτό που είπα εγώ προκαταρτικά βέβαια είναι διαταπερισμένος ο χώρος αυτός ε, της έκθεσης γιατί δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ένα κάποιο όγκο αλλά υπάρχει διάθεση σε αυτά που ζητούν οι συνάδελφοι. Ε, το συμφωνώ μαζί και τώρα Τσίλτερ ε, η συνάδελφος μιλάει για την καλύτερη πρόσβαση για τις ε, υπηρεσίες της υγειονομικές και για την Ευρωπαϊκό Χάρτη Κινητικότητας. Είναι σημαντικά αυτά τα σημεία και εγώ τα βρίσκω σημαντικά και θα τα δούμε αυτά μαζί τις μέρες τις επόμενες Στάφος Ότζες, ναι, να υπάρξει μια συμπλήρωση, το συμμερίζομαι αυτό και ταυτόχρονα από τη στιγμή που θα ε, υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση, διαφορετικά θα μπορούσαν να το παραμελήσουν αρκετά κράτη-μέλη. Ενώ από τη στιγμή που θα υπάρξει ένα κονδύλι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν αρκετοί. Και η εκπαίδευση, κατάρτιση είναι κάτι το σημαντικό γιατί κάτι τέτοιο επιτρέπει μια ευκολότερη ένταξη στο χώρο εργασία και το σχέδιο μείωση τη φτώχεια για κατοικία, εξέβρεση κλπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που φεύγει από το σπίτι οικογένειά του, το άτομο αυτό με προβλήματα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα για να ενταχθεί στην κοινωνία και η εκστρατεία επίση ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντική για εκείνου που δεν έχουν παρόμοια προβλήματα, αλλά θα πρέπει να κατονίσουν τα προβλήματα των άλλων. Ε, Χουμπνερ, ναι, για την πρόσβαση αυτή, όχι μόνο ε, για το πρώτο σκέλος αλλά και για τις υπηρεσίες και θα πρέπει όχι μόνο να τους βοηθήσουμε όταν θα πρέπει να πάνε σε ένα γραφείο, σε ένα οργανισμό και στο νοσοκομείο αλλά στο σύνολο της ζωής τους, στη διασκέδασή τους, στον σε αθλήματα παντού και από τη στιγμή που θα ενταχθεί η κοινωνική πρόνοια ε, είναι το, το καταληκτικό, το τελευταίο γιατί εκείνος που έχει προβλήματα έχει δικαίωμα να ζει καλύτερα. Άρα λοιπόν εδώ έχει δικαίωμα για κάτι παραπάνω. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Σαν Πρόντι, ναι, για την ε, ενημέρωση είναι κάτι το σημαντικό και αυτό το έχω εντάξει εγώ. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες ενημέρωσης, πληροφόρησης, ώστε και τα άτομα με ιδιαίτερες αναπηρίες και μεγάλα προβλήματα να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και διάφορες υπηρεσίες για καλύτερη ποιότητα ζωής. Επίσης να ευχαριστήσω την Επίτροπη η οποία προχώρησε σε μια ανακοίνωση την οποία πλήρως συμμερίζομαι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο τη μερισσιακή διάταξη και περνάμε στο επόμενο σημείο. Ή μάλλον να μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα τη έκθεση ρωση Ρώση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 3η Μαΐου. Έγκριση στην Επιτροπή μα στι 24 Μαου και στην Επιτροπή Απασχόληση στι 16 Ιουνίου. Και τώρα ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της διάταξης. Άρα, περνάμε στο επόμενο. Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για μια έκθεση πρωτοβουλία Επιτροπής ΙΤΡΕ. Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα. Θα δώσω το λόγο στην συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Βάνα Πλάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.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 να δώσω συγχαρτήρια στην Επιτροπή βέβαια η οποία δημοσίευσε μια ανακοίνωση για τις προτεραιότητες για την δομή την ενεργειακή για την ε, πριν και την μετά το 2020 περίοδο. Και στην γνωμοδότησή μου εγώ προσπάθησα να τονίσω διάφορες πτυχές πάνω απ' όλα τις ε, επενδύσεις που απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές σε αυτό στην Ευρώπη από τη στιγμή που θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους που επιδιώκουμε. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρθηκε ένα απαραίτητο ποσό 200 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε στο δίκτυο να εντάξουμε τις νέες τεχνολογίες και να μπορέσει να επεκταθεί επίσης η υποδομή μας στο σύνολό της. Θα πρέπει στα πλαίσια αυτής της χρηματοδότησης να κατανοήσουμε ότι αν δεν γίνουν με σωστό τρόπο τότε θα μας κοστίσει ακόμα περισσότερο επειδή θα χειροτερεύσει η κατάσταση ε, και στο περιβάλλον και επειδή θα έχουμε μια εξάρτηση ψηλότερη, μεγαλύτερη όσον αφορά την ενέργεια. Για να μην μιλάμε τώρα και για τη μείωση της ευμάρειας αλλά και τη μείωση των θέσεων εργασίας. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι τα ταμεία αυτά θα πρέπει να υποστηριχθούν και να έχουν ε, δημόσια κονδύλια και ιδιωτικά κονδύλια και για τα δημόσια κονδύλια εδώ θα πρέπει να πρόκειται ας πούμε για τους φόρους ε, για το διοξείδιο του άνθρακος κλπ. Με αυτές τις δημόσιες επενδύσεις θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους υπόλοιπους και για περαιτέρω επενδύσεις από ιδιωτικής πλευράς σύμφωνα με τις ανάγκες ε, και τη ζήτηση που υπάρχει και τη χρησιμοποίηση ε, πηγών ενέργειας πράσινες. Κάτι που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι χρειάζεται να αποφύγουμε, να παρακάμψουμε τους κινδύνους ε, που είναι και φυσικοί κίνδυνοι αλλά και οφείλονται σε εμά τους ίδιους και στην πολιτική που ασκούμε και το κόστος και το όφελος θα πρέπει να καταμετρηθούν και στα πλαίσια της οδηγίας του 2008 πάνω στις κρίσιμες φύσεως υποδομές. Και επίσης οι επενδύσεις χρειάζεται να καταλάβουν σε εισαγωγικά ότι υπάρχουν αυτές, αυτοί οι κίνδυνοι. Θα ήθελα να υποδείξω στα κράτη-μέλη να χαράξουν ένα χάρτη, ένα χάρτη που θα μας δείξει πώς έχει κατάσταση και πώς, τι γίνεται με τις μέχρι τώρα υπάρχουσες επενδύσεις αλλά να λάβουμε υπόψη μας και τους κινδύνους επαλαμβάνω που μπορούμε και πρέπει να παρακάμψουμε και το πώς θα συνδυάσουμε τα διάφορα εθνικά δίκτυα. Επίσης, από τα κράτη-μέλη ζητάω να δώσουν στους πολίτες, στην κοινωνία των πολιτών, τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν και στους οικονομικούς φορείς, όπως επίσης και στους κοινωνικούς εταίρους, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε νέες ενέργειες και μάλιστα με έξυπνο τρόπο που να είναι και αποτελεσματικές. Κάτι ακόμα ότι απαιτεί το εξυγχρονισμό των εθνικών δικτύων ενέργειας και επίσης ένα υπερδίκτυο έξυπνο με μια σταθερή ροή ενέργειας με προσιτές τιμές για τους πολίτες έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πολλών θέσεων εργασίας και μάλιστα πράσινες θέσεις εργασίας. Να τονίσω επίσης ότι οι πολίτες χρειάζεται να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Και ειδικά ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν προτεραιότητα τα σχέδια εκείνα, τα προγράμματα εκείνη που απασχολούν περισσότερο από τα υπόλοιπα τους πολίτες. Τους κοιόδης συγητές να τους ευχαριστήσω, όπως και τη γραμματεία της Επιτροπής που επέτρεψαν την ε, οργάνωση μιας ανεπίσημης συνάντησης στο Στρασβούργο για το θέμα αυτό. Τους ευχαριστώ. Περιμένω δε τις σκέψεις, τις απόψεις, τις ιδέες των ε, συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ, Χιούμπνερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Η εισηγήτρια έθεσε αρκετά ζητήματα στην γνωμοδότησή της και νομίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση για αυτό το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2007 ενέκρινε σημαντικούς στόχους ε, για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της ανταγωνιστικότητας, της σταθερότητας ε, και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Το 20% πρέπει να, της ενέργειας πρέπει να πρόκειται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επίσης πρέπει να μειωθούν κατά 20% εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να αυξηθεί επίσης κατά 20% η ενεργειακή απόδοση. Όμως η συγκεκριά έχει εστιάσει στην περιβαλλοντική πολιτική, στην πολιτική για το κλίμα, για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εσγασίας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και στην ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, γιατί αυτό είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Εξίσου σημαντική είναι η ίση πρόσβαση στην αγορά ενέργειας. Διότι ο χρόνος ζωής των επενδύσεων στον τομέα αυτό ο χρονικός ορίζοντας, αν θέλετε, είναι πολύ μεγάλος, είναι πολύ μακρύς. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε όλοι οι αποδέκτες ε, της ενέργειας, ε, βιομηχανίες και νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν αυτή την ενέργεια. Επενδύσεις. Επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αυτό ζητείται να συμπεριληφθεί στον οδικό χάρτη για το 2050. Θα υπάρξει σχετική δημοσίευση φέτος στο φθινόπωρο, αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να δεχόμαστε λύσεις που δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί ως προτεραιότητες από το Συμβούλιο. Άρα δεν μπορούμε εμείς να προβαίνουμε σε τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες είναι πρόορες. Σε ό,τι αφορά το εδάφιο 4, ναι, υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλεία. Συμφωνώ. Πρέπει να είναι ορθολογικά αυτά τα πρότυπα και να αποσυνδεθούν από άλλες παραμέτρους, ανάπτυξη υποδομών ή διασύνδεση των δικτύων. Διότι αυτές οι συνδέσεις δεν υλοποιούνται γιατί υπάρχει συχνά αντίσταση για τέτοιου είδους έργα. Θα πρέπει λοιπόν τα πρότυπα ασφαλείας να είναι λογικά και να μην εμποδίζουν τη διασύνδεση μεταξύ δικτύων. Πρέπει να είμαστε λογικοί και πρέπει να βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα. Εδάφιο 5. Γίνεται λόγος εδώ για την αποθήκευση, αποθήκευση του ηλεκτρισμού. Είναι όπως ε, εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, ένα πρώιμο στάδιο της επιστημονικής έρευνας αυτό και δεν έχουμε ακόμη τεχνολογίες που να προβλέπουν την αποθήκευση χωρίς μείωση της απόδοσης. Ή τεχνολοποτέλεσμα τελικά να μειώνεται η απόδοση με αυτήν την ε, αποθήκευση του ηλεκτρισμού. Τώρα, ανανεώσιμες πηγές σε σχέση και σύνδεση με τα δίκτυα. Δεν μπορούμε αυτή, σε αυτό το στάδιο να πραγματοποιήσουμε το στόχο αυτό, εάν δεν εντοπίσουμε, αν δεν βρούμε ποιος είναι ο, ο ιδιοκτήτης του δικτύου που θα πρέπει να προβεί σε, αυτό το, σε αυτή τη διασύνδεση και να φτιάξει αυτό τον κόμβο διασύνδεσης. Το κόστος μιας τέτοιας διασύνδεσης δεν θα πρέπει να το φέρουν ε, οι πελάτες ε, οι ε, ιδιώτες. Θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα που, ποιον βαρύνει το κόστος αυτό. Εδάφιο 7. Αναφέρεται μια εξαιρετική πρόταση της Επιτροπής. Να έχουμε ένα γενικό πρόγραμμα, για κάποια προγράμματα προτεραιότητας. Έργα προτεραιότητας και για αυτά θα πρέπει να έχουμε ταχύτερες και διαφανέστερες διαδικασίες έκδοσης άδεια. Και βέβαια γίνεται λόγος για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων. Αυτό που λείπει όμως είναι η ενημέρωση, η πληροφόρηση του κοινού. Και εκεί ε, δημιουργούνται προβλήματα για την ε, λειτουργία ορισμένων από αυτές τις υποδομές. Άρα είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται αυτή η ενημέρωση στον πληθυσμό, στο κοινό και αυτό να γίνεται αρκετά νωρίς. Όχι να περιμένουν να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα έργα αυτά, γιατί τότε θα είναι αργά. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε περισσότερους μέσα από αυτές τις πτυχές. γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, θα αυξηθούν. Και πάλι όμως η προσέγγιση μας πρέπει να είναι ισορροπημένη. Και αυτές οι πηγές ενέργειας θα πρέπει να διασυνδεθούν σωστά στο δίκτυο παροχής ενέργειας. Ιδίως όταν μιλάμε για διεθνές δίκτυο ενέργειας, ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς αποτελεσματικά αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κυρία Βίλς από τη ΓΟΕ σας ευχαριστώ πολύ. Λέει η κυρία Βίλς. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Πλουμ. Στο Στρασβούργο είχαμε ήδη την ευκαιρία να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων για το θέμα αυτό και εγώ πιστεύω ότι και οι στόχοι κατά πολέμηση κλιματικής αλλαγής και οι θέσεις εργασίας που έχουν πράσινο χαρακτήρα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θέλω να τονίσω και μερικά ακόμα σημεία τα οποία με ενδιαφέρουν προσωπικά. Καταρχήν, η ανάπτυξη μια υποδομή ενέργεια για τι ανανεώσιμε ενέργειε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επιτύχουμε. Και όταν μιλάμε για ανανεώσιμες ενέργειες, μιλάμε επίσης και για αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας. Δεν θέλουμε να έχουμε όμως περισσότερες υποδομές για τον άνθρακα, για την πυρηνική ενέργεια, για τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας θα πρέπει εν καιρό, μακροπρόθεσμα τουλάχιστον, να εγκαταλείψουμε την πυρηνική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο είναι η άποψή μου ότι οι υποδομές ενέργειας θα πρέπει να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης, γιατί αλλιώς αν το αφήσουμε αυτό στα χέρια των εταιριών, οι εταιρείε ουσιαστικά τα μετακυλίουν στους καταναλωτές και καθορίζουν τα δίκτυα όπως θέλουν αυτοί. Εμείς θέλουμε στη Γερμανία να γίνει πάλι δημοτικοποίηση, να αναλάβουν οι δήμοι την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα της απλοποίησης, της αδειοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται με ταχύτερο τρόπο η αδειοδότηση και να μην υπάρχει τόσο μεγάλο άχθος, τόσο πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια για αυτούς που υποβάλλουν ε, αιτήσει προς την κατεύθυνση αυτή και θα πρέπει να υπάρξει και μια δημόσια συμμετοχή στις διαδικασίες έγκρισης κατασκευής δικτύων ή σταθμών ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να γίνεται με πιο γρήγορο ρυθμό όταν υπάρχει και πλήρης ε, εμπλοκή των ενδιαφερομένων και του πληθυσμού, γιατί αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να καταθέτουν και εναλλακτικέ τάσεις, ώστε να υπάρξει λοιπόν η διαδικασία διαμόρφωσης μια άποψης που θα κάνει το σχέδιο αυτό αποδεκτό για τους τοπικούς κατοίκους. Αυτό θα είναι υπέρ της διαδικασίας και θα μειώσει τις αντιδράσεις. Επίσης θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της ε, αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας <clears throat> γιατί με καλύτερες υποδομές μπορούμε να επιτύχουμε και μορφές εξοικονόμησης ενέργειας και καλύτερης αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας. Και για να επιτύχουμε λοιπόν τους στόχους αυτούς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και τα δίκτυα διανομής για τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες και για την αποκεντρωμένη κατανομή της ενέργειας, τα δίκτυα αυτά να μπορέσουν να τελειοποιηθούν και να συμπληρωθούν, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξει και ανταλλαγή ενεργείας μεταξύ κρατών μελών και μετακίνηση ενέργειας με εύκολο τρόπο, χωρίς ε, απόλυση. Κύριε Κωνσταντς, Γκροστέτ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ, όταν πρόκειται για παρόμοιες ε, δομές για το 2020 το χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε σε μεγάλες επενδύσεις. 200 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη δεκαετία για να αποκριθούμε στις ανάγκες. Ε, οποιοδήποτε και είναι ο τρόπος ε, παραγωγής ενέργειας. Χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Χρειαζόμαστε την οργάνωση, την υποδομή αυτή. Τώρα η σημερινή οικονομική κρίση ίσως και αποτελεί την ευκαιρία να δούμε κάποιες αναλυτικές λύσεις στη σημερινή κατάσταση με καινοτομίε τεχνολογικές και με την έρευνα μια παρότριση και με πηγές ανάπτυξης και επίσης περισσότερες θέσεις Γι' αυτό χρειάζεται την κοινοτομία και την έρευνα να την υποστηρίξουμε και επίσης να έχουμε μια ενεργού πολιτική χρηματοδότησης με καινοτόμα μέσα και εργαλεία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, επίσης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα υπάρχοντα κονδύλια και τα βιέ, ε, χρηματοδότηση και καλύτερη κατανομή των ε, ε, κονδυλίων, να δούμε ακριβώς και τα ιδιωτικά γεγονότα που συμμετάχουν, αφού θα κάνουμε μια εκτίμηση των κινδύνων και επίσης ένα δασμό, ένα φόρο για την πράσινη ενέργεια και για τον άνθρακα και τα διάφορα άλλα συστήματα και όλα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν με κονδύλια σε αυτή τη χρηματοδότηση. Την υποδομή μας λοιπόν απόλυτα θα πρέπει να την προσαρμόσουμε στον δικό χαρακτήρα αυτό της μεταφοράς παρόμοιας ενέργειας και να εντάξουμε γίνεται καλύτερα αυτό τον δικό χαρακτήρα για την ε, ολική ηλιακή ενέργεια γιατί ακριβώς έχουμε ένα, ένα σύστημα που δείχνουμε ότι διαφοροποιείται αυτή ε, η βεντάλια η πλατιά. Και επίσης να μειώσουμε την ε, ενεργειακή εξάρτηση, περισσότερη αποτελεσματικότητα ενεργειακή, ανταγωνιστικότητα καλύτερη από πλευράς ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας, κυρίως των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων και έτσι να μπορέσουμε να ελέγχουμε καλύτερα, να καλύτερα την ενεργειακή μας κατανάλωση και στο τέλος θα έχουμε κέρδο οικονομικό αλλά και πάνω στο περιβάλλον. Αυτά λοιπόν είναι τα κάποια λίγα που θα ήθελα να προσθέσω στην έκθεση αυτή και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέω Κύριος Όντι είναι ο, ο επόμενος Πρόντι συγκεκριμένα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τη συνάδελφα Πλάμ θα ήθελα να την ευχαριστήσω και να τη συγχαρώ για την έκθεσή της γιατί είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Να πω μερικά πράγματα συγκεκριμένα για διάφορα θέματα που μάλλον θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε σχέση και με τα καινούργια που μας είπε η Επιτροπή την ανακοίνωσή της. Γι' αυτό ναι, αυτός ο δικός χάρτης της Επιτροπής για το 2050 μήπως αυτό θα σημάνει και μια κάποια αλλαγή, μεταβολή σε σχέση με τις υπόλοιπες προθεσμίες όπως του 2020. 2020, εντάξει για το 2020. Νομίζω ότι αποτελεί κάτι το σημαντικό το οποίο σίγουρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Να προσθέσω και κάτι άλλο. σε σχέση πάντα με την έκθεση αυτή. Τι παρατηρώ. Ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον για κάποιες πτύχες, μία συστηματική προσέγγιση ολική και ανάμεσα στην ανάγκη που παρουσιάζεται για μια προσαρμογή που έχει σχέση με το κλίμα, την αλλαγή του κλίματος που έχει ήδη σημειωθεί και που χρειάζεται μια ειδική συμπεριφορά, ας την πούμε σε εισαγωγικά διατήρηση εδώ του χώρου ας πούμε, κάτι που κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, αλλά θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν από τη στιγμή που με συστηματικό τρόπο θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε είδους ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που υπάρχει επί τόπου. Και μάλιστα μιλώντας ειδικό για την βιομάζα και τα απόβλητα, τα γεωργικά, τα δασικά επίσης και ακόμη για το πώς θα διατηρηθούν οι δατινοί πόροι, ποτάμια, ριάκια και υπόλοιπα και πώς θα, αυτά θα τα βελτιώσουμε, πώς θα τα βοηθήσουμε και πώς με υδραυλικά μέσα εκτός από το να προσφέρουμε ενέργεια μέσω αυτής της δραυλικής ε, εκμετάλλευσης θα μπορούσαμε να προσέξουμε και το περιβάλλον παράλληλα και ταυτόχρονα. Να λοιπόν, ε, αυτές οι συνθήκες ε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την κλιματική αλλαγή και να εγγυθούμε και μια προσαρμογή του χώρου, του περιβάλλοντος, του εδάφους ε, σε αυτό το πρόβλημα που το θεωρούμε θεμελιώδους σημασία και σας ευχαριστώ βέβαια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως η εισηγήτρια, λέει η κυρία Βάλεαν, στην Επιτροπή Βιομηχανίας τόνισα τη σημασία να επενδύσουμε στα FEE e δίκτυα διανομής νομίζω ότι είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες μας. Χαίρομαι που ο εισηγητής, η εισηγήτρια συγκεκριμένα, υπογράμμισε το σημείο αυτό σε πολλές παραγράφεις. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε <clears throat> την ε, πλήρη ολοκλήρωση των νέων ενεργειών στα δίκτυά μας προς όφελος των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες ενέργειες, θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι αυτός είναι ο δρόμος, ένα τμήμα του δρόμου του μέλλοντος. Δεν πρέπει να βλέπουμε όμως την κατάσταση σε μαύρο ή σε άσπρο μονάχα. Και οι τεχνολογίες οι ανανεώσιμες έχουν επίπτωση και στο περιβάλλον. Όταν αποφασίσουμε πού επενδύουμε και πώς επενδύουμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό τον παράγοντα και θα λάβουμε υπόψη και το κόστος το οποίο έχει να κάνει με την ε, ε, εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών. Έχουμε δει τις προτάσεις της Κομισιόν και τα αριθμητικά στοιχεία που μας έδωσε ότι υπάρχει αυξανόμενη, αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και ανάγκη εξυγχρονισμού των υποδομών. Εγώ είμαι μια φιλελεύθερος και εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ένα φόρο ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών για τη χρηματοδότηση των αναγκών μας. Η εισηγήτρια λοιπόν δεν θα πρέπει να εντάξει αυτή την ιδέα στην γνωμοδότησή της και να ξεκινήσει μια εκστρατεία για αυτό το θέμα, ένα θέμα για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιτύχει ευρύ βαθμό συνένεσης. Θα πρέπει αντίθετα να είμαστε δημιουργικοί και να βρούμε νέα εργαλεία λαμβάνοντας υπόψη την τωρινή οικονομική κατάσταση και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα λεγόμενα project bonds σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η αγορά θα πρέπει να οδηγεί. Οι επενδύσεις της αγοράς θα πρέπει να είναι αυτές οι οποίες θα έχουν την πρωτοκαθεδρία, εκτός της περιπτώσεις που δεν υπάρχει κίνητρο για εμπορικές επενδύσεις. Τότε μπορεί να λάβει τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα project bonds της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ο κυριότερος μοχλός για την επιτυχία, <clears throat> για την ε, εγκαθίδρυση αυτών των υποδομών που χρειάζονται όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά και για τις μεταφορές και για άλλους χώρους. Τέλος, συγχαίρω την συγκίτρια για το δύσκολο έργο που έφερε σε πέρας και ελπίζω θα συνεχίσουμε την συνεργασία μέχρι το αίσιο πέρας αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε Λίζερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πλόμπα, την συγκίτρια Θα ήθελα να σταθώ σε ένα στοιχείο αυτής της συζήτησης και θα προετοιμάσω και τροπολογίες σχετικά. Είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε υποδομές και χρειαζόμαστε και ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε όμως και τα πράγματα από την οπτική γωνία του καταναλωτή. Έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη αποδοτικότητα της ενέργειας. Αν δούμε λοιπόν το πώς θα μειώσουμε την ε, κατανάλωση ενέργειας σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθεί η χρήση ενέργειας. Γι' αυτό η Κομισιόν ώψη του 2020 και του 2050 θα πρέπει να έχουν ρεαλιστικές προβλέψεις για την ε, ζήτηση από τους καταναλωτές θα είναι πολύ πιο χρήσιμο να δώσουμε έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και όχι μόνο στην αύξηση των ανανεωσίμων ενεργειών και θα πρέπει να σκεφτούμε και για μια καλύτερη διαχείριση της ζήτησης. Έχουμε πολλές φορές ενέργειες οι οποίες έχουν διακειμενόμενη παροχή στο δίκτυο <clears throat> και αυτό θα μας, πρέπει να μας οδηγήσει να καταλάβουμε καλύτερα πότε χρησιμοποιεί ο καταναλωτής το δίκτυο ενέργειες και πότε όχι. Πολλές φορές έχουμε παραδείγματος χάρη εγκαταστάσεις ψήξεως οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την τροφοδοσία με ενέργεια σε σταθερό επίπεδο. Αν τώρα έχουμε όμως ε, τροφοδοσία μονάχα με ανεμογεννήτριες, άμα δεν λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες λόγω ελήψεως ανέμου, τότε το ψυγείο αυτό, οι εγκαταστάσεις ψήξης, θα έχουν μονάχα μία ώρα περιθώριο αποθηκευμένη ενέργεια μέχρι να μείνουν από ενέργεια. Επομένως θα πρέπει να έχουμε μια γενικότερη αντιμετώπιση για τις ανάγκες σε ενέργεια και θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα και για τα αυτοκίνητα και την αυτοκίνηση. Τα αυτοκίνητα <clears throat> ουσιαστικά κυκλοφορούν δύο ώρες την ημέρα και κάθονται 22 ώρες την ημέρα. Αν βρούμε ένα σύστημα ε, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να τροφοδοτούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όταν υπάρχει περισσεύον ρεύμα με φτηνό τρόπο, αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει και τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά φυσικά, να δρούν ως αποθήκες ηλεκτρικής ενέργειας και μπορούν και τα αυτοκίνητα μετά όταν κινούνται να αποδίδουν ενέργεια σε άλλες χρήσεις ενέργειας. Επομένως δεν πρέπει να σκεφτούμε μονάχα την ευφυά <clears throat> ανάπτυξη δικτύων ως ε, τρόπο αντιμετώπισης της ε, ζήτησης ενέργειας, αλλά ως τρόπο ολοκληρωμένης διαχείρισης της ενέργειας. Το τελευταίο σημείο, η χρηματοδότηση εδώ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Όλοι ε, δεν είμαστε, διστάζουμε να πούμε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τους καταναλωτές στο δίκτυο, αλλά υπάρχει και η αρχή του ότι ο χρήστης πρέπει να έχει την ευθύνη. Εφόσον, εφόσον οι καταναλωτές αυτοί που χρησιμοποιούν τα δίκτυα, αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος αυτό. Τώρα όταν πρόκειται για αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ περιορισμένη ε, χρήση δικτύων, αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι η ΕΤΕΦΑΟ, παραδείγματος χάρη η Γερμανία ή άλλες, αυτές ουσιαστικά αποκομίζουν το κέρδος τους από την ιδιοκτησία που έχουν τα δίκτυα. Επομένως θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι όποιος θέλει να αναπτύξει τα δίκτυα θα πρέπει αυτός να τα χρηματοδοτήσει. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να σκεφτούμε ποια είναι η καλύτερη λύση από ευρωπαϊκή και από εθνική πλευρά για την χρηματοδότηση αυτών των δικτύων. Ευχαριστώ. <clears throat> Σας ευχαριστώ. Πάλι ο λόγος στην συγκήτρια. Και νομίζω ότι και ο κύριος Πρόντι είχε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα για την Κομισιόν η οποία απουσιάζει σήμερα. Αλλά οι υπηρεσίες μας θα τις εκμεύσουν απαντήσεις στα ερωτήματά σας και δεν έχω ακούσει τώρα άλλα ερωτήματα από συναδέλφους προς την Κομισιόν, αλλά αν έχετε συγκεντρώστε τα για να τα υποβάλουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Δίνω και πάλι το λόγο στην κυρία Πλόμπ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τις ε, συνεισφορές τους. Δυστυχώς ξέρετε ότι οι διαδικασίες μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω μονάχα 1500 χαρακτήρες. Γι' αυτό δεν, μπορέ, δεν να επεκταθώ στο βαθμό που θα ήθελα σε αυτή τη γνωμοδότηση. Θα οργανώσω και πάλι μια συνάντηση με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους για να συζητήσουμε για τις τροπολογίες. Τώρα δεν θέλω να δώσω μια απάντηση σε όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν. Αλλά Σίγουρα θα έχουμε με την συμβολή σας μια πολύ καλή έκθεση η οποία ως υπόψη τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την διαχείριση ενέργειας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει και ηγέτης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και να γίνει ένα σημαντικό παίκτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των σημαντικών κλιματικών και ενεργειακών θεμάτων. Και επίση για την ασφάλεια, για την υγεία και την οικονομική ασφάλεια όλων των πολιτών της Ευρώπης. Θέλω και γι' αυτό τον λόγο να σας ευχαριστήσω και θα ξανασυζητήσουμε για τις συγκεκριμένες τροπολογίες που θα υποβάλλετε. Σας ευχαριστώ τα μάλα. Thank you Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. <clears throat> Το προσωρινό χρονοδιάγραμμα προβλέπει προθεσμία κατάθεση τροπολογιών μέχρι τι 2 Μαου. ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας 24 Μαου και στην Επιτροπή Ήτρε στις 26 Μαΐου και η έκθεση στη συνέχεια θα έρθει τον Ιούλιο στο, στην Ολομέλεια. Κλείνουμε αυτό το σημείο της μέσης διάταξης λοιπόν και περνάμε στο επόμενο που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Κομισιόν, την ε, Υπηρεσία Φαρμάκων και άλλους φορείς για το αντιδιαβητικό φάρμακο Mediator. Και ξεκινάμε δίνοντο το λόγο στους εκπροσώπους της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα για να πατήσουμε στην ερώτηση για το Μετιατόρ. Εισαγωγικά να πω κάποια πράγματα. you know, started, you know, in... Η όλη υπόθεση ξεκίνησε το 1999. Προποντού υπάρξει νομοθεσία για τη φάρμακο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εισήχθη το 2004 για πρώτη φορά και συγκεκριμένα περιλαμβάνει κανόνε περί φαρμακοεπαγρύπνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνέχεια αυτή η νομοθεσία ενισχύθηκε το 2010, πρόσφατα δηλαδή. Το φαινόμενο πέρυσι εγκρίθηκε αυτή η νέα νομοθεσία. Η νέα νομοθεσία, ξέρετε, ενισχύει, ξέρετε, το ρόλο της φαρμακοεπαγρύπνησης που ξέρετε ότι θέλουμε να τονίσουμε. Την εποχή του Μεντιατόρ υπήρχε ομάδα εργασίας. Αυτό πλέον έχει γίνει, θα γίνει επίσημα επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης τώρα. Και με τη νέα νομοθεσία έχουμε τη διαχείριση των κινδύνων των φαρμάκων ε, που διευρύνεται. Δηλαδή η ερμηνεία του τι εστί κίνδυνος, ξέρετε, τώρα διευρύνεται και περιλαμβάνει και τα λεγόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Επίσης υπάρχει πλέον η δυνατότητα, ξέρετε, να περιληφθεί στην έγκριση, στην άδεια κυκλοφορία ενός φαρμάκου, ε, διάταξη και όρος ε, για την παρακολούθηση. Όταν ε, προέκυψε το θέμα με το Mediator, μας συζητήθηκε να κάνουμε μια δοκιμή αντοχής, ένα stress test, για να δούμε κατά πόσον σήμερα με την νέα νομοθεσία τη δομοσία του 2010 που θα τεθεί σε ισχύ του χρόνου αν το Μεντιατόρ θα ξανασυνέβαινε. Και πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς ε, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι ότι ναι, θα ξανασυνέβαινε ίσως αντίστοιχη περίπτωση Μεντιατόρ. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί και η νομοθεσία μας. Πρόκειται βέβαια για νομοθεσία που μόλις εγκρίθηκε και όπως είπα θα τεθεί σε ισχύ του χρόνου. Η ανάλυση μας όμως ξέρετε λέει ότι αν θέλουμε να είμαστε 100% σίγουροι δεν θα ξαναέχουμε περίπτωση σαν το Μεντεατόρ στο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την νομοθεσία. Και υπάρχουν τρία κυρίως θέματα επί των οποίων η νομοθεσία μας δεν είναι ακόμη αρκετή. Τα εξής. Πρώτα απ' όλα, όταν υπάρχει εθνική απόσυρση, πάντοτε πρέπει να ξεκινούν κοινοτικές διαδικασίες. Στην περίπτωση του ξέρετε, ξέρετε, δεν υπήρξε, ξέρετε, ποτέ εθνική απόσυρση. Ξέρετε ότι δεν έγινε τέλος πάντων αυτή η απόσυρση δυστυχώς, αλλά ακόμη και αν είχε γίνει, ξέρετε, δεν υπήρχε υποχρέωση για το κράτος μέλος ε, να φέρει το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό για μας αποτελεί εγγύηση γιατί έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ε, που είναι ο θεματοφύλακας και έχουμε και αυτή την Επιτροπή για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση τώρα. Δεύτερον, υπάρχουν εταιρείε φαρμακευτικές που αποσύρουν εθελοντικά κάποια φάρμακα. Θυμάστε τι έγινε με το Mediator. Το 99 Ιταλία και Ισπανία σταμάτησαν να διαθέτουν στο εμπόριο το φάρμακο αυτό γιατί ε, η εταιρεία το απέσυρε θελοντικά. Δεν υπήρχε όμως υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών. Γιατί, γιατί έγινε αυτό. Γιατί η εταιρεία δηλαδή απέσυρε το προϊόν σε κάποια κράτη-μέλη συγκεκριμένα. Άρα, όταν υπάρχει θελούσια, θελοντική απόσταση του φαρμάκου, τότε πρέπει υποχρεωτικά η εταιρεία να ενημερώνει τι αρχέ και να δικαιολογεί την απόσταση, να δίνει τους λόγους για τους οποίους το αποσύρει. Αν λοιπόν η Εθνική και η Ευρωπαϊκή Αρχή γνωρίζουν γιατί υπάρχει απόσταση, αυτό είναι σημαντικό. Τρίτον, νομίζουμε ότι η ανάγκη για διαφάνεια σε όλες αυτές τις έρευνες μετά την ε, κυκλοφορία των ε, φαρμάκων είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Δηλαδή τώρα έχουμε βάση, θα έχουμε βάση δεδομένων και θα συλλέγουμε όλα τα δεδομένα από τις μελέτες post-monitoring. Και τα δεδομένα όλων αυτών των μελετών μετά τη διάθεση του φαρμάκου στο εμπόριο θα πηγαίνουν σε μια βάση δεδομένων. Έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα υπάρχει υποχρέωση σε αυτή τη βάση δεδομένων να την Έτρανετ όπω λέγεται, να μπαίνουν εκεί όλα τα στοιχεία από τις μελέτε μετά την ε, κυκλοφορία του φαρμάκου, μετά την έγκρισή του. Σε νομοθετικό επίπεδο πρέπει να γίνει, όπως ξέρετε, όπως είπα, και άλλη δουλειά. Η υπόθεση του Μεντιατόρ δημιουργήθηκε και έγινε γιατί τότε υπήρχε εθνική αρμοδιότητα, δεν υπήρχε ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, δεν υπήρχε αρμοδιότητα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Νομίζουμε τώρα ότι ο Οργανισμός Φαρμάκων και η Κομισιόν έδρασαν ε, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες. Και τώρα, επαναλαμβάνω, υπάρχει η ευρωπαϊκή αρμοδότητα. Ευχαριστώ πολύ. E να δώσω το, τον λόγο στον κύριο Αντρέα Σπότα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να πάρω θέση για την περίπτωση Mediator Ben Fluorex. όπως έχει λεχθεί, ούτε η Κομισιόν ούτε ο Οργανισμός Φαρμάκων έχουν κάποια άμεση ευθύνη. Είχαν κάποια άμεση ευθύνη για το προϊόν αυτά και την ομάδα προϊόντων αυτών. Από το 1998 στο 2000 είχαμε συζητήσει για το θέμα αυτό στην λεγόμενη ομάδα φάρμακο επαγρύπνησης. Θα επανέλθω τώρα για το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων. Υπήρξαν ορισμένες προειδοποίησης αλλά δεν διαπιστώθηκε με άμεσο τρόπο η τοξικότητα αυτού του προϊόντος. Υπήρξαν προειδοποίησεις οι οποίες οδήγησαν στην απόσυρση του φαρμάκου αυτού από την Ιταλία. Στο χρονικό διάστημα 2000 με 2009 ο Οργανισμός Φαρμάκων δεν αντιμετώπισε καθόλου το φάρμακο αυτό. Μόνο από το 2009 έγινε το, ε, υπήρξε το πρόβλημα αυτό με το Fluorex και στη συνέχεια αποσύρθηκε από την αγορά. Δεν είχαμε καμία λοιπόν ευθύνη για το φάρμακο αυτό στα αρχικά ε, επίπεδα. Το θέμα αυτό συζητήθηκε μονάχα στα πλαίσια της ομάδος φάρμακο επαγρύπνησης που έχει, σας πεντιμίζω, δύο λειτουργίες. Μία ευρωπαϊκή λειτουργία και μία διακυβερνητική λειτουργία. Η ευρωπαϊκή λειτουργία αφορά προϊόντα τα οποία μέσω της, ε, του Οργανισμού Φαρμάκων και της Κομισιόν την χάνουν ε, κεντρικής έγκρισης. Ήταν τότε 120 προϊόντα του 1998, τώρα είναι πάνω από 600, αλλά υπάρχουν πάνω από 90.000 προϊόντα τα οποία την χάνουν εθνικής έγκρισης και για τα οποία έχουν απόλυτη αρμοδιότητα τα εθνικά, οι εθνικές αρχές. Γυρίστε τώρα στο 1998. Ήταν μια κούτσικη μικρή υπηρεσία η, η ΕΜΕΑ, ο Οργανισμός Φαρμάκων και έπρεπε να αγωνιστεί για να μπορέσει να βρει τη θέση της έναντι των ισχυρών, των πανισχύρων εθνικών αρχών έγκρισης για τα φάρμακα. Μέσα στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε η ομάδα εργασίας για την φάρμακοεπαγρύπνηση, η οποία θέλησε να αναπτύξει κάποιες ευρωπαϊκές διαδικασίες αλλά οι εκπρόσωποι των κρατών μελών <clears throat> εξακολουθούν να <clears throat> συζητούν εκεί για τα εθνικά τους προϊόντα και μετά μπαίνουν στην, γυρίζουν στη χώρα τους και εκεί ακολουθούν τις εθνικές αρχές έγκρισης. Λοιπόν δεν ήταν το αγαπημένο παιδί κανενός ο οργανισμός φαρμάκων αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα στην αρχή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι μήπως θα έπρεπε αυτό το προϊόν να το αναλάβει ο οργανισμός φαρμάκων. Ακόμα και στο διάδρομο και στο καφενείο δεν μπορούσαμε να τολμήσουμε να πούμε κάτι τέτοιο. Μπορείτε να φανταστείτε ένα τέτοιο οργανισμό ο οποίος επί τρία χρόνια δεν είχε τη δυνατότητα να πει τίποτα ούτε στους Γάλλους ούτε στους Ιταλούς είτε σε κανέναν άλλο ότι τα προϊόντα σας είναι επικίνδυνα γιατί έτσι θα έπαβε να υπάρχει πια αυτός ο οργανισμός φαρμάκων. Επομένως υπήρξε ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο δεν έδωσε καμία δυνατότητα για την ΕΜΕΑ, και τον Οργανισμό Φαρμάκων, να προχωρήσει σε ρύθμιση για ορισμένα φάρμακα. Η φορέα φαρμάκων μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τα φάρμακα τα οποία βρίσκονται στη δική του αρμοδιότητα. Αλλά δεν μπορεί να δεχτεί ότι για τα προϊόντα ε, που υπόκειται στην επικουρικότητα και επομένω στι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ζητηθούν ευθύνες από τον Οργανισμό Φαρμάκων. Εάν υπάρξει μια νέα νομοθεσία, θα μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη αρμοδιότητα στα θέματα αυτά, αλλά μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Φάρμακα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στι εθνικέ αρμοδιότητε. Κύριε Σένμαρη, ίσως θα θέλατε να λάβετε το λόγο και να παρουσιάσετε τον εαυτό σας για το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μέρος της Γενικής Επιθεώρησης Κοινωνικών Υποθέσεων, ακριβώς το Σώμα Επιθεωρητών, στην υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας. Πρώτη φορά που λαμβάνω το λόγο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν ξέρω εάν ε, γνωρίζω την ορολογία που απαιτείται, συγγνώμη πάντως, και θα ήθελα να συμπληρώσω από τη στιγμή που συμφωνείτε τα λόγια του συναδέλφου μου, του προηγούμενου που έλαβε το λόγο, να αναπτύξω δύο σημεία. Εμείς αυτό που δείξαμε τώρα δεν είναι κατά την απόψή μας θέμα ρύθμισης και το δεύτερο να προσφέρουμε συγκεκριμένα στοιχεία τι γίνεται στην Ευρώπη για τον Μπενφλόρεξ. Να πούμε κάτι για το πρώτο σημείο. Τι είδαμε, τι παρατηρήσαμε. Είναι καταστροφή υγειονομική για την υγεία στη χώρα μου και ασχολείται η δικαιοσύνη, έχει επιληφθεί του θέματος. Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα ρύθμισης, και υπάρχουν διάφορα κενά τα οποία πλήρως έχουν περιγραφεί λίγο πριν. Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο σημεία επίσης σε θέματα ρύθμισης. Μπορεί να υπάρχει μια κάποια ρύθμιση, αλλά ίσως δεν εφαρμόζεται κατάλληλα και δεν υπάρχουν και κυρώσεις. Είχαμε αρκετές περιπτώσεις αυτά τα τελευταία τελευταία χρόνια για το Μεντιάτορ ας πούμε που δεν εφαρμόστηκε αυτός ο κανονισμός και δεν υπήρξαν κυρώσεις και να επιμείνω σε κάτι ότι ε, στα φάρμακα έχουμε να κάνουμε με μια ρύθμιση που είναι τρόμερα σημαντική. 10.000 ρυθμίσεις διάφορες και θα μπορούσα να σας πω μερικά πράγματα για αυτά, για τα φάρμακα ακριβώς. Είσαι 100.000 ε, φάρμακα διπλασιάστηκαν μετά τα τελευταία δέκα χρόνια που μετά από τον τρόπο μας οδήγησαν σε πολλές νομικές πτυχέ και δεν υπάρχει όμω κατάλληλη προτεραιότητα εκεί που πρέπει έτσι θολά κάπω ε, ασχολούμεθα όχι με την πανεκτίμηση των υπαρχόντων και ε, για να δείξουμε το υπάρχει και τη χρήση και για το μεντιατόρο υπήρχε το 70% το συνταγών, συνταγογράφησης, χωρίς όμως την εξοδότησή της θέσης του προϊόντος στην αγορά. Εδώ να σας πω, αυτό ήθελα να σας υπενθυμίσω ακριβώς και κάτι ακόμα που παρατηρήσαμε στην έρευνα αυτή. Είχαμε και προβλήματα ρυθμίσεων αλλά υπήρχαν και κενά του οργανικού φορέα. Είχαν να κάνουν ε, με τη ρύθμιση σε διαφορετικά τρία σημεία οργάνωση, μέθοδο και γενική αντιμετώπιση για την οργάνωση τώρα. Υπήρχε ιδιαίτερο φόρτο εργασία, ε, κάποιο που λαμβάνει χιλιάδε αποφάσει το χρόνο, οργάνωση περίπλοκη με 2.000 εμπειρογνώμε, φαρμακοεπαγρύπνηση εδώ, με διάφορου παράγοντε που ασχολούνται και με το κόστο όφελο, ε, κίνδυνο, ε, φαρμακο που έχει να κάνει και με πολλή δουλειά και εκεί ασχολούνται πάντα όλοι αυτοί οι μυρογνώμονες του συμφέρει να απασχολούνται επί μακρόν. Αυτά λοιπόν. Έχουμε διάφορε εθνικέ ομάδε εργασίας, οι οποίες όμως ε, ε, δεν είχαν μια κάποια πίξη σωστή φαρμακολογικά και ούτε την, ε, τα πραγματική ζωή, τι συμβαίνει καθημερινά όσον αφορά τα φάρμακα και δεν εκτίμησαν όπως πρέπει αυτές τις παρενέργειες. Επίσης, δεν έλαβαν υπόψη τους ε, τα ανησυχητικά σήματα από την Ιταλία και την Ισπανία και πάντα τι προσπαθούσαν επιστημονικά με την εταιρεία να τα βρουν και υπήρχαμε και 35 μελέτες για το Mediator και ε, με πάμπολε σελίδε καταλαβαίνετε και ακόμα κάτι προσέξτε στο τέλος τέλος είναι και μία θέμα συνήθειας οι συνήθειες μας οι νομικο έχουν σαν επίκεντρο αυτό το φάρμακο και ε, ο φορέας το μερίζεται με τις φαρμακευτικές εταιρείες και για το όλο ε, περιεχόμενο αυτορυθμίσεων και επειδή ξέρουμε ποιο είναι το κείμενο, είναι το φάρμακο και η αντίληψή μας δεν έχει να κάνει κυρίως με το πώς μέσω του φαρμάκου θα περίσσουμε σε μια στρατηγική θεραπευτική που να βασίζεται στον ίδιο τον παθόντα, τον ασθενή και δεν είμαστε και τόσο ανοιχτοί σε κάτι άλλο από την άλλη μεριά, μάλλον ε, και αντιμετωπίζουμε αυτά που λένε ε, οι υπόλοιποι, γιατί είναι το κράτος, είναι οι ασθενείς, όλοι αυτοί ρύθμισαν το πρόβλημα τελικά, ε, το πρόβλημα του Μεντιτάτορ στη Γαλλία και όχι ο φορέας κλπ. Και επίσης μια κάποια αμφιβολία που είναι υπέρ όμως του φαρμακού και μια προληπτική μέθοδος που είναι υπέρ του φαρμάκου και όχι υπέρ του ασθενούς. Τώρα, σε λίγα λεπτά επιτρέψτε μου να πω μερικά πράγματα για το τι έγινε από το 1998 μέχρι το 2003. Το 1998 η Ιταλία, ο καθηγητής Γκαρατίνη, που είναι ξέχουσα φυσιογνωμία και κάποιος ακόμα από το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας, οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό και κάλεσαν τον Ευρωπαϊκό Φορέα ακριβώς για το θέμα του Mediator και η Ιταλία με τη βοήθεια της Γαλλίας συντάσσει μια έκθεση ιδιαίτερα συγκεκριμένη, περιληπτική, ακριβή και που λέει τα εξής. Ε, δεν είναι σχεδόν καθόλου αποτελεσματικό το φαρμακό αυτό. Και ακόμα υπάρχουν ε, παρενέργειες, ε, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, ιδιαίτερες παρενέργειες και ακόμα χημικά μοιάζει πολύ αυτό το προϊόν ε, με τα φάρμακα κατά της ανορεξίας, ε, καταλαβαίνετε. Αλλά δεν παρακολουθεί και το θέμα ως πρέπει. Και η έκθεση της Ιταλίας έλεγε ότι θα πρέπει να ζητηθεί μια διατησία βάσει του άρθρου 12 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής, δηλαδή να ζητήσουμε μια επανεκτίμηση του ωφέλους και του κινδύνου. Και αυτή η διατησία δεν ζητήθηκε ποτέ ούτε από την Ιταλία ούτε από τη Γαλλία. Τώρα η Ιταλία τι υποστηρίζει. Χρειάζεται μια καινούρια, χρειάζονται καινούργιες ε, εκθέσεις ε, για την καρδιοτοξικότητα ας πούμε του προϊόντος από τα εργαστήρια τα και ε, κατέληξαν μετά από δέκα μήνες συζήτηση για μια μελέτη αλλά δεν πραγματοποιηθεί κανείς δεν θα την πραγματοποιήσει ε, τόσο καιρό μετά έγινε και μια καρδιογράφημα κάπως στο τέλος ε, που βλέπουμε ότι βάσει αυτών κατηγορείται όμως το φάρμακο αυτό και επίσης υπάρχει έκθεση ιταλική που λέει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για να συμπεριλάβουμε τους κινδύνους καρδιοτοξικότητας και η Γαλλία ε, δεν θα το αλλάξει και όπως είπαν οι συνάδελφοι, το 2003-2004 ε, η ίδια εταιρεία από την Ισπανία και στην Ιταλία αποσύρει το φάρμακο και βλέπουμε τι έγινε από γαλλικής πλευράς μέχρι το 2009 όμως. Αυτά, αυτά θα ήθελα να αναφέρω εδώ μπροστά στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι συνάδελφοι οι οποίοι θα θέλανε να λάβουν το λόγο. Η κυρία Γκρός Τέτς έχει το λόγο καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή την πολύ ατυχή υπόθεση που συζητάμε έχει διάφορες επιπτώσεις. Εδώ εμπλέκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός Φαρμάκων, και ο, η ε, συντάξη έκθεσης ε, για το φορέα το γαλλικό ΙΓΚΑΣ, προσπαθούμε όλοι αυτοί να βρουν τις ε, συνέπειες και τις ευθύνες που υπάρχουν και είναι πολλαπλές. Δεν είναι ενός μόνο η ευθύνη, υπάρχει αλυσίδα ολόκληρη ευθυνών με αμέλειες, πολύ σοβαρές και είναι γεγονός ότι πρέπει να ενισχύσουμε οπωσδήποτε η νομοθεσία μας. Πρέπει να πω ότι οι συνθήκες ήταν πρόσφαρες διότι τον Νοέμβριο του 2010 ψηφίσαμε την αναθεώρηση, την ενίσχυση της φαρμακοεπαγρύπνησης. Βέβαια, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Επιτρόπο Πονταλή, αμέσως μετά από την ε, δρομολόγηση αυτών των stress test, αφού επιλήφθηκε του θέματος ο Επίτροπος, είδαμε ότι υπάρχουν τρία δυνατά σημεία, τα εξήγησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην αναθεώρηση νομοθεσία του 2010 σε σχέση με τι είχαμε ψηφίσει το 2004. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής ε, νομοθεσίας το 2004 και θυμάμαι πολύ καλά τις συζητήσει που είχαμε τότε. Πράγματι, όταν η Γαλλία ζήτησε ή μάλλον αποφάσισε την αναστολή ε, του Μεντιατόρ το 2009, αυτό είχε γενική επίπτωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί είχαμε την εφαρμογή της νομοθεσίας το 2004 και τελικά με τη νέα νομοθεσία το 2010 αυτό δεν θα είχε γίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν και σωστά ο Επίτροπος ε, Νταλή έκανε αυτή τη δοκιμή αντοχής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αδυναμίες και τις εξήγησε πάρα πολύ ωραία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το ερώτημα που θέλω εγώ να θέσω τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη στιγμή που Έγινε η διαπίστωση αυτή. Πώς τώρα θα τροποποιήσουμε την νομοθεσία. Πώς μπορούμε να το κάνουμε. Ο Επίτροπος Νταλή το Μάιο θα πρέπει να μας κάνει πρόταση για την ενημέρωση των ασθενών. Και είναι σημαντικό πολύ γρήγορα να μπορέσουμε αυτές τις σκέψεις να τις ε, εντάξουμε πως και τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής και να είμαστε έτσι πιο αποτελεσματικοί. Όπως υπόθηκε, δυστυχώς έτσι είναι οι άνθρωποι, ε, το σφάλιν ανθρώπινων και ποτέ δεν θα ε, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος ε, να ξανασυμβεί μια τέτοια υπόθεση, αλλά πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οποτεδήποτε υπάρχει τέτοια υποψία να μπορούμε να έχουμε τις σωστές αντιδράσεις. Θέτω λοιπόν στην Κομισιόν αυτό το ερώτημα. Τι μπορούμε να υποθέσουμε, τι μπορεί να προβλέψει ο Επίτροπος Ντάλι για το θέμα αυτό. Τώρα, είναι γεγονός ότι η νομοθεσία, η ρύθμιση δεν τα προέβλεπε όλα. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να σκεφτούμε και ποια θέση θα έχουμε για την ε, χορήγηση φαρμάκων εντός αδειών ε, κυκλοφορίας. Ακούω αυτά που μας λέει ο κύριος Σέτιεν Μαρή. Το 2004 ήμουν συγκίτρια, Εγώ σα είπα για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα φάρμακα. Εγώ τότε ήθελα να περνάμε από ευρωπαϊκές άδειες κυκλοφορίας σε και αν αυτό γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από όλα τα κράτη-μέλη, άρα δεν υπάρχει διάκριση σε βάρος κάποιων Ευρωπαίων πολιτών, και αν υπάρξει αναστολή να είναι γενική και άμεση αυτή η αναστολή τη κυκλοφορία του φαρμάκου. Και τότε δεν θα είχαμε το πρόβλημα τη Γαλλία που περίμενε μέχρι το 2009 για να αναστείλει αυτή, την κυκλοφορία αυτού του φαρμάκου. Αυτό το οποίο λέω και επαναλαμβάνω και ξαναλέω είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δίνονται ώστε να το περισσότερο κυκλοφορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ενισχύεται η πεποίθησή μου όταν ακούω αυτά που μου λέει Μαρή. Δηλαδή, αν ε, υπήρξαν όλα αυτά τα προβλήματα, οι ανεπάρκειες, οι αμέλειες από τον αρμόδιο γαλλικό φορέα, ήταν γιατί είναι βεβαρημένος με πάρα πολύ έργο. Και δεν μπορούσε να τα προλάβει όλα. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι τα όρια Ε, και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει τι άδειε κυκλοφορία των φαρμάκων να τι δίνει το συντομότερο δυνατό πλέον ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Φάρμακων. Θα μου πείτε, ναι, θέλετε να μειώσετε του εθνικού οργανισμού φαρμάκων, τι θα του κάνουν, πώ θα του χρηματοδοτήσουμε, θέλουν να έχουν κάποια έσοδα. Ναι, πράγματι υπάρχουν προβλήματα πραγματικά και πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Τουλάχιστον έχουμε αυτή τη θετική πλευρά. Υπάρχει και ένα ερώτημα που θέλω να θέσω στον κύριο Ετιέν Μαρή Στη Γαλλία είχαμε πάρα πολλές εξεταστικές επιτροπές ε, εξε, την, ε, από την Εθνοσυνέλευση, από την ε, Γερουσία, το ΙΓΚΑΣ, είχαμε κάποιο κογκρέσο για την εξόρυξη των φαρμάκων, Φιλίπ Εβά. όλα αυτά, πάρα πολλές εκθέσεις και μπορώ να αναφέρω και πολλές άλλες εκθέσεις και εξεταστικές επιτροπές και δημιουργείται σύγχυση. Κυρίως όμως τελικά λησμονούμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στη Γαλλία Τίνουμε να το ξεχνάμε αυτό. Ας αρχίσουμε λοιπόν να εφαρμόζουμε καλά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί μόλις έγινε αναθεώρηση φαρμακοεπαγρύπνησης, πλέον είναι ανάγκη να γίνει μεταφορά αυτών των διατάξεων στο εθνικό δίκαιο. Α το κάνουμε πλέον γρήγορα στη Γαλλία για μια φορά, να είμαστε σύμφωνοι λοιπόν με αυτήν την νομοθεσία. Ο κύριο Ντάλι θα μα κάνει προτάσει από πλευρά κομισιών για την ενημέρωση των ασθενών Ας βιαστούμε λοιπόν στην Γαλλία να μεταφέρουμε γρήγορα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δίκαιο ε, ώστε να έχουμε λιγότερα προβλήματα. Κύριε Τιεν Μαρή, σας ερωτώ, έχετε υπόψη συνεχώς ότι δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε γαλλογαλλικά τα πράγματα, αλλά να εργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί έχουμε πολύ καλή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω, γιατί νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Νομίζω ότι γρήγορα τα είπα, αλλά είχα να πω και τόσα πολλά. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά ένα σκάνδαλο εδώ που έπληξε πολλούς ε, Γάλλους και Γαλλίτες αλλά και πολλούς άλλους Ευρωπαίους που ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους ως συνέπεια του προβλήματος αυτού, διότι οι υπεύθυνοι δεν πήραν τις σωστές πολιτικές αποφάσεις για το θέμα αυτό. Εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι οποίοι όπως πολύ σωστά το υπογράμμισε η κυρία Γκροστέτ έχουμε θεσπίσει νομοθετικές ρυθμίσεις για την φαρμακοεπαγρύπνηση τόσο το 2004 όσο και το 2010 το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να επιτύχουμε την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της νομοθεσίας για να αποφευθούν παρόμοια προβλήματα. Εμείς είμαστε στην Επιτροπή η οποία ασχολείται ακριβώς με αυτά τα προβλήματα υγείας. Και αντίθετα από αυτά που μας είπε ο Επίτροπος Νταλή, απαντώντας σε ένα προφορικό ερώτημα που του είχα θέσει 15 Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια του Στασβούργου, δεν πρόκειται εδώ και το είπατε και εσείς κυρία μου, δεν πρόκειται και μόνο για ένα πρόβλημα που αφορά τη Γαλλία. Παρά το γεγονός ότι από το 2005 λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα εργαστήρια Σερβιέ είχαν αποσύρει εθελοντικά το φάρμακο αυτό και από την Ιταλία και από την Ισπανία, το φάρμακο αυτό κυκλοφορούσε μονάχα στη Γαλλία. Και εξάλλου από την άλλη πλευρά η γαλλική δικαιοσύνη έχει να φέρει σε πέρα στο έργο της και θα διαπιστώσει ενδεχομένω ποινικέ ευθύνε. Όχι, πρόκειται όμω για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, όπω πολύ σωστά είπατε, γιατί θα έπρεπε εμεί όλα αυτά τα χρόνια να πράξει τα αναγκαία ώστε ο Ευρωπαϊκό Φορέα για τα Φάρμακα, ο ΕΜΕΑ, να έχει τι απαραίτητε δομέ φαρμακοεπαγρύπνηση και έγκαιρη προειδοποίηση για να πει στι εθνικέ αρχές ότι ένα φάρμακο θα πρέπει να απαγορευτεί μετά από αυτά που έλαβαν χώρα σε μια άλλη χώρα μέλη. Μέλος είναι απαραίτητο πάντα να υπενθυμίσω ότι εμείς δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Και εσείς βέβαια από την υπηρεσία φαρμάκων το είπατε ότι δεν υπήρχε η νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορέσει να το κάνει αυτό ο φορέας φαρμάκων. Αλλά αν θέλαμε να φτάσουμε στο τέλος θα έπρεπε όλοι να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι ακούγοντα αυτά που είπε όχι μόνο η εκπρόσωπο της Κομισιόν αλλά και τους δύο άλλους παρεμβαίνοντες. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο μας πρότεινε ο Επίτροπος, ε, Νταλή μέσα στα πλαίσια μιας ε, παραδοξότητος ίσως λέγοντας ότι είναι ένα γαλογαλικό πρόβλημα αλλά θα το χρησιμοποιήσω και στα, τέσσερα αντοχή στο Νομίζω ότι με αυτά που είπατε κυρία εκπρόσωπε της Κομισιόν, το πρόβλημα αυτό ήταν πραγματικά ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να μπορούμε να αποτρέψουμε στο μέλλον τέτοια προβλήματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει εκ βάθρων η νομοθεσία στα θέματα αυτά. Όπως ελέγχθη και το 2004 και το 2010 έγιναν αλλαγές, αλλά αυτό δεν είναι επαρκές. Δεν αρκεί να έχουμε νέες οδηγίες για την πληροφόρηση των ε, ασθενών. Όχι. Είναι το σύνολο του συστήματος το οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί. Γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να πράξουμε τα απαραίτητα για να γίνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις για το σύστημα φάρμακο επαγρύπνησης για να σταματήσουν αυτές οι συγκρούσεις συμφερόντων που εμποδίζουν την αποτελεσματική ρύθμιση στον τομέα των φαρμάκων. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε κάνει είτε το 2004 είτε το 2010 στον τομέα αυτό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση που εγκρίναμε το 2010, ναι μεν προχωρεί προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα <clears throat> για τις εγκρίσεις θέσεις σε αγορά των προϊόντων θα έπρεπε η ευρωπαϊκή διαδικασία για την ε, ε, έγκριση των φαρμάκων θα έπρεπε να δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν περισσότερο μηχανισμοί της αγοράς και να υπάρχει και ένας ευγενής ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών για να επιτύχουν μια καλύτερη αναγνώριση των προϊόντων τους. Αυτό θα έπρεπε λοιπόν να είχε γίνει. Οι εθνικές αρχές όμως προσπαθούν πάντα να βρούνε με ένα μέσο δρόμο μεταξύ των αναγκών εξασφάλισης δημόσιας υγείας και της θέλησης να προσελκύσουν τις μεγάλες εταιρείε. Προς το συμφέρον λοιπόν ε, του Ευρωπαίου καταναλωτή και πολίτη είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας κώδικας καλής δεοντολογίας και συμπεριφοράς από την πλευρά όλων των εμπλεκομένων στην αδειοδότηση των φαρμάκων. Όπως είπατε κυρία μου, από την Κομισιόν έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα των τεστ αντοχής τα οποία έχουν γίνει, αιτήσει του Αρμοδίου Επιτρόπου και πιστεύω ότι θα έχουμε το σύνολο αυτών των συμπερασμάτων όσον ούπο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα συμπεράσματα για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνουμε μια μικρή μονάχα τροποποίηση στην οδηγία για την πληροφόρηση των πολιτών, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για μια πλήρη αναδιάταξη του συστήματος και των κωδικών, των κωδίκων συμπεριφοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για μένα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Αφού διάβασα όλες τις προφορές, έχω σχηματίσει και την προσωπική μου άποψη Παρ' όλα αυτά, εμάς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να πρόκειται να λάβουμε μια σοβαρή απόφαση και όταν νομοθετούμε βάση βέλτιστων πρακτικών αυτό δεν μας απαγορεύει από το να νομοθετούμε και βάση κάποιων κακών πρακτικών. Δεν είναι γαλλογαλλική υπόθεση, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παράδειγμα και είναι ένα επιχείρημα για την ανασφάλεια δικαίου, τα κενά, τη γραφειοκρατία, πάρα πολύ πολύπλοκες διαδικασίες, όλα αυτά ε, και συμφωνούμε με το Συμβούλιο, ε, δημιουργούν πολύπλοκες διαδικασίες, ε, κάποιες φορές εξυπηρετώντα φέροντα το κλάδο, αλλά ε, δημιουργούν προβλήματα για το δημόσιο συμφέρον. Και πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα έχουμε σαφή στοιχεία γιατί ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα. Υπήρξε μια αντίφαση και διαφωνία μεταξύ εθνικών φορέων και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Και τελικά υπήρξε η νομοθεσία να έχει μεγαλύτερη εξουσίες και αρμοδιότητε ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά το Συμβούλιο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι ικανοποιημένο με όλε τι προτάσει, οποίε εμεί ω Κοινοβούλιο προσπαθούμε να προωθήσουμε με την νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνηση και το Συμβούλιο εξακολουθεί να απορρίπτει ορισμένε από τι προτάσει μα και ιδίω αυτέ που σχετίζονται με τη διαφάνεια. Να σας θυμίσω όταν ε, έγινε μια πρόταση εδώ στο Κοινοβούλιο για την ε, αποκάλυψη, την κοινολόγηση συγκρόσεων συμφερόντων υπερογνωμόνων ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, καταψηφίστηκε αυτή η πρόταση και αυτό με εξέπληξε και εμένα και όλους όσους ήμασταν υπέρ αυτής της πρότασης. Εννέα ψήφταν διαφορά δεν πέρασε η πρόταση και το επιχείρημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ήταν ότι είναι πάρα πολύ πολύ τελικά και θα δημιουργήσει διοικητικό άχθο για του υπεργονόμενου αν θα πρέπει να κάνουν δηλώσει σύγκρουση συμφερόντων και να ε, αποκαλύπτουν τέτοιε περιπτώσει. Μιλάμε για 10% άτομα και κάθε φορά έχουμε εδώ πέρα 2.000 ε, συνεργάτες οι οποίοι υπογράφουν αυτές τις δηλώσεις σύγκρουση συμφερόντων. Δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν, που όμως εδώ μπορούν να είναι επικίνδυνα και για το κοινό. Λοιπόν, τρεις συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να αποτρέψουμε. Πρώτον, εθνική σύγκρουση συμφερόντων. Και έχουμε στο γαλλογαλλικό πρόβλημα. Πράγματι, εδώ έχουμε εθνική σύγκρουση συμφερόντων. Σε βάρος του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Έχουμε εθνικό προστατευτισμό. Μετά, πολιτική σύγκρουση συμφερόντων. Υποθέτω όμως ότι τα γαλλικά δικαστήρια θα το ξεκαθαρίσουν αυτό και όλοι όσοι ενέχονταν ιδρύματα, φορείς, οργανισμοί, και όπως όλη αυτή η διαδικασία προχωρεί. Και μετά έχουμε, όπως είπα, την Εθνική Σύγκρουση Συμφερόντων. Έχουμε τώρα έρευνα η οποία χρηματοδοτείται, επιδοτείται από τη βιομηχανία, από τον κλάδο. Στην περίπτωση φαρμάκων από τη Merck και την Pfizer. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε και πόσο οι αποφάσεις μας και οι οργανισμοί μας είναι αξιόπιστοι. Είχαμε μια απόφαση πρόσφατα της ΕΦΣΑ για την ασφάλεια των τροφίμων που αφορά κάποιες αξιώσεις για την υγεία στον δομέα των τροφίμων. Είχαμε έρευνα που πρότεινε, έκανε κάποιες αξιώσεις για την υγεία για το βρεφικό γάλα και θέλαμε επιστημονικά στοιχεία από πανεπιστήμια, από ανεξάρτητες αρχές. Αυτά τα στοιχεία ήταν κατά αυτών που υποστήριζε η βιομηχανία, που υποστήριζε ο κλάδος. Και εμείς είπαμε, εμείς εμπιστευόμαστε την ΕΦΣΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλισης των Τροφίμων. Αλλά πώς μπορούμε να επισκεφθούμε αν δεν έχουμε μια σαφή ε, δήλωση περί μη σύγκρουση συμφερόντων και αν μπορούμε να έχουμε τελικά εμπιστοσύνη σε αυτούς τους οργανισμούς και αυτούς τους φορείς. Φυσικά και υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας περί φαρμακοεπαγρύπνησης και αναμένω τη νέα πρόταση του κυρίου Νταλή, του Επιτρόπου, το Μάιο. Διότι ο Επίτροπο πολύ ξεκάθαρα είπε ότι δεσμεύεται να επιβάλλει μεγαλύτερη διαφάνεια και αποκάλυψη ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή τέλο πάντων αποτροπή περιπτώσεων σύγκρουση συμφερόντων για αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με την δημόσια ασφάλεια και υγεία. Να συμπληρώσω ότι εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε πολλά παραδείγματα όταν ψηφίζουμε δηλαδή δεν ψηφίζουμε πάντοτε υπέρ ε, ή προς το συμφέρον τη κοινή γνώμη. Γι' αυτό λοιπόν ε, ζητώ ότι πρέπει και εμεί να δείξουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και σοφροσύνη. Για να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να πανερχόμαστε, να υπαναχωρούμε και να ξαναεξετάζουμε την νομοθεσία μα. Και τέλο να πω ότι αυτή δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε η πρώτη ούτε η μοναδική περίπτωση για τη μη μεταφορά τη κοινοτική νομοθεσία στη Γαλλία και όχι μόνο και σε άλλα κράτη-μέλη. Έχουμε τρει οδηγίε σε σχέση με τα μοσχεύματα που δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Τώρα έχουμε τη φαρμακοεπαγρύπνηση που δημιουργεί ζήτημα και έχει να κάνει και με το τους πίνακες σε αυτό που το βλέπουμε κάθε φορά. Και με το Συμβουλίο θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά γιατί τα 9-10 χρόνια που είχαμε αυτή την υπόθεση πέθαναν δύο-τρει χιλιάδε άνθρωποι. Αυτό είναι το τίμημα λοιπόν αυτή τη ανασφάλεια και αυτή τη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συνάντηση αυτή με όλους ε, από την Ούγκα στη Γαλλία τον επιθεωρητή και την Επιτροπή ε, και ανησυχώ, ανησυχώ πάρα πολύ για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Τώρα σε τι εξυπηρετεί αυτός ο φορέας, τι γίνεται. Το 1999 είχαμε την έκθεση Ιταλίας, ζήτησε μια διαιτησία για να δει ακριβώς ε, το κόστος ε, κίνδυνος. Τι έκανε ο φορέας αυτός. Τίποτα. Το 1999 είπε το ΕΜΕΑ, Α, εγώ δεν διέθετα για να ενεργήσω την κατάλληλη νομική βάση, την νομοθεσία. Και μετά το κοφάν ε, προτείνει να το αποσύρει αλλά για το Μεντιάτορο δεν λέει τίποτα. Ενώ η φεμφλουραμίνοι ακριβώς προκαλούσε ανορεξία και μάλιστα σε υψηλό βαθμό, ήταν επικίνδυνο. Λοιπόν, ενώ άλλο φάρμακο το απέσυρε. Γιατί δεν το έκανε το ίδιο με το Μεντιάτορο. Και στο Άφσα, στη Γαλλία, ο επικεφαλής ε, και στο ΕΜΕΑ, ποιος είναι ο επικεφαλής, ο Ζαμπιερ Αλεξάνδρα, που είναι από τη Γαλλία με τον Αποδαράκη και με, ασχολείται με την φαρμακοεπαγρύπνηση ε, στον, ευρωπαϊκό, στον φορέα αυτό, στο ΕΜΕΑ. Εδώ μην ξεχνάμε ότι του κυρίου Γκαρατίνη η έκθεση ήταν ιδιαίτερα σαφή συγκεκριμένη. Έλεγαν στα εργαστήρα Σερβιέ να διεξάγουν μία μελέτη που είχε μεγάλη σημασία για τις ε, καρδιακές παρενέργειες. Και τι έγινε το 2006 πια εννέα χρόνια μετά έχουμε ένα φάρμακο που δημιουργεί πρόβλημα και κανείς δεν προχωράει σε αυτή την μελέτη. Τι κάνετε εκεί εσείς αυτό το φορέα σας. Και μετά έχουμε τον Ρίκ Καμπαντή, ο οποίος ακολουθεί τη δουλειά αυτή, είναι στο γαλλικό φορέα διευθυντής και από την άλλη μεριά έχει ορισμένες, ε, μια υπεύθυνη θέση στην ε, φαρμακοεπαγρύπνηση. Ένας Γάλλος σε αυτές τις δύο θέσεις πάντα. Τι γίνεται λοιπόν. Εδώ έχω αυτήν την επιστολή. Το 2000 ε, χτυπάει το καμένο κινδύνου η Ισπανία και λέει ακούστε αυτό το φάρμακο το Mediator χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ε, σαν ανορξιογόνο ε, και όχι για το διαβήτη. Για πέστε μας τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Το 2004 έχουμε ακόμα μια επιστολή που ε, ναι, αντίθετα με αυτό που λέτε εσείς κύριε μου από την Επιτροπή ενημερωθήκαμε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στα ΜΕΑ και αναφερόταν υπάρχει πρόβλημα, πρόσεξε και πάλι τα εργαστήρα Σερβιέ αποσύρουν το φάρμακο αυτό τι κάνει το MA. Και από τους Γάλλους, από τους Ιταλούς το βλέπω αυτό το 2003. Τι κάνει ο φορέας, τίποτα αυτός ο εξοργασμός φαρμακών. Και πρέπει το 2006 επιτέλους ε, να κάνει μια μελέτη, μια μελέτη και τότε να διαπιστωθούν αυτά τα καρδιακά προβλήματα. Τι κάνει αυτός ο εξοργασμός φαρμακών. Θα πρέπει να περιμένουμε, είχαμε την Ερενφεσό που είναι πνευμονιολόγος, ο οποίος γιατρός ακριβώς και λέει προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε στην αγερμός, καρδιοπάθειες. Και μετά τον Ιούνιο του 2010 επιτέλους ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου ε, αποφασίζει την απόσυρση του φαρμάκου. Τι να σας πω τώρα εγώ αποκαρδιωμένη. Εντάξει, εξοδοτήσει και λοιπά ευρωπαϊκές. Εγώ εντάξει δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτό. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Εσείς τι κάνατε. Εντάξει, στη Γαλλία σχέσεις με τα... Σιωπή, <laughs> κυρία Φωστέτ, εγώ σα άφησα να μιλήσετε. Λοιπόν, ε, ανάμεσα στα εργαστήρια Σερβία και τους εμπειρογνώμονε, μια συνεργασία κτλ. Τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά στην Ευρώπη τι γίνεται, δεν το καταλάβατε το συναγερμό αυτό, με αφού ορισμένα κράτη σα λένε ότι υπάρχουν καρδιοπάθειες που σημειώνονται ακριβώ λόγω της χρήσης του φαρμάκου αυτού, της λήψη του φαρμάκου αυτού. Τι γίνεται, γιατί κανείς δεν το βλέπει αυτό. Το πάντεριξ επίση. Ε, υπήρξε μια άδεια για το πάντεριξ από το GSK τα εργαστήρια αυτά και πρώτη συναγερμό που χτύπησε από τους Σουηδού, λέτε τα παιδιά που παίρνουν το πάντεριξ έχουν ε, εννέα φορές περισσότερα προβλήματα ε, για προβλήματα ναρκοληψίας και καταλαβαίνετε ακριβώς και οι Σουηδικές αρχές είπαν ότι το Μεμρίξ αποσύρεται ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα υπνηλίας ε, και ακόμα ε, μετά τι γίνεται παρόλο στις παραπάνω φορές κινδύνου και τι κάνει το Παεμρίξ λέει δεν το αποσύρω ακόμα έρευνες τι γίνεται πόσους νεκρούς περιμένετε πρώτα πόσοι πρέπει να πεθάνουν για να ξεκινήσει η όλη πορεία και η έρευνα είναι ιδιαίτερα δίνει η περίπτωση απέναντι στην περίπτωση απέναντι εδώ απέναντι στους επιθεωρητές εάν αυτός ο οργανισμός φαρμάκων είναι εκεί ακριβώς για να λέει το ναι, δηλαδή το πράσινο φως στα φάρμακα και μια χρηματοδότηση 90% από τι εταιρείε φαρμάκων και δεν προσέχετε του ασθενεί, αλλά προσέχετε αντίθετα τα εργαστήρια, τα φαρμακολογικά, καταλαβαίνετε, τα φαρμακευτικά, καταλαβαίνετε είναι άσχημη κατάσταση. Παρακαλώ, διαβάσετε την έκθεση Λίγκας. Κάθε φορά λέτε ότι εδώ πώς εμπλέκεται ε, η κατάσταση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, γιατί, γιατί ε, δεν παίρνουν εκεί μέτρα, περίμενα την Ευρώπη να τα λάβει. Τι έγινε, ο διευθυντής τι λέει, α, δεν είχαμε στα χέρια μας τα την απαραίτητη νομοθεσία. Ναι, αλλά για τον ρεξιογόνα το κάνατε αυτό πράγμα. Τι κάνατε, ε, τα διάφορα εργαστήρια όταν από εδώ και από εκεί σε κάθε κράτος σας λένε προσέξτε, συναγερμός κίνδυνο και εσείς αδιαφορείτε. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί η φαρμακοπρεκρίνηση αν είναι εσόφλος των ε, ε, φαρμακευτικών εταιριών τότε εγώ ανησυχώ τι κάνει τότε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Κυρία Ροτ Μπέραντ, σας ευχαριστώ. Ίσως χρειάζεται κάποια περισσότερη ηρεμία σε αυτή τη συζήτηση και μια καλύτερη οργάνωση και διάρθρωση της συζήτησης. Καταρχήν, ο καθένα ο οποίο έχει την εντύπωση ότι, ότι με την τροποποίηση τη νομοθεσία για τη φάρμακο επαγρύπνηση, είτε είναι χρήσιμη είτε δεν είναι χρήσιμη αυτή η αλλαγή, ότι με αυτή την περίπτωση, ότι με την αλλαγή τη νομοθεσία μπορεί να αποτρέψει μια περίπτωση όπω αυτή του Mediator, αυτό είναι σφάλμα τελείω. Όσο υπάρχουν ακόμα οι εθνικές αδειοδοτήσεις, εφόσον επιτρέπουμε να υπάρχουν εθνικές αδειοδοτήσεις θα υπάρχουν πάντα τέτοια φαινόμενα. Όπως είπε και η Φρανσουάζ, ε, εγώ πάντα υποστήριξα την ευρωπαϊκή αδειοδοτήσεις. Όλοι θέλαν και οι Γάλλοι όμως και οι Γερμανοί και όλοι θέλουν να κρατήσουν την εθνική αδειοδότηση. Γιατί υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα αυτό και όλοι θέλουν να τους διατηρήσουν στις θέσεις εργασίας τους. Και όταν εγώ λέω, κυρία Ριβάση, να έχουμε μια ευρωπαϊκή αδειοδότηση, όταν την έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή αδειοδότηση, τότε μπορείτε να φωνάζετε όσο θέλετε. Γιατί δεν έχει γίνει όμως αυτό το πράγμα. Το καθεστώς της ΕΜΕΑ, γιατί όπως όλοι οι αποκεντρωμένοι φορείς έχει ένα καταστατικό, το καταστατικό ήδη του φορέα φαρμάκων καταδεικνύει και ποιες είναι οι αρμοδιότητες Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το καταστατικό αν θέλουμε. Γιατί αυτό προβλέπει όπως και σε όλους τους αποκεντρωμένους φορείς τι μπορεί να κάνει. Και το ίδιο γίνεται και με την ΕΦΣΑ, με την εταιρεία, την υπηρεσία για την τροφιμική ασφάλεια. Υπάρχουν σε όλες αυτές τις ε, υπηρεσίες σαφής δομής. Αλλά τα κράτη-μέλη δεν θέλησαν τα τελευταία 15 χρόνια να υπάρχει αυτός ο Ευρωπαϊκός Φορέας για τα φάρμακα. Το είπε ο πρόσωπο της ΕΜΕΑ. Τα κράτη-μέλη δεν το θέλησαν να υπάρχει αυτό το σύστημα. Και εξασφαλίσαν να υπάρχει στην Επιτροπή αυτών των φορέων και ένας εκπρόσωπος από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, κοιτάξτε το αυτό κύριε Αριβάζη. Εγώ είμαι η πρώτη η οποία θα ήθελε να καταργηθεί αυτό το σύστημα. Αλλά πρέπει να αλλάξετε προηγουμένως το καταστατικό αυτών των φορέων. Ότι κάθε κράτος μέλος έχει τον ε, μπάστακά τους αυτούς τους φορείς. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος από τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Πρέπει να το δούμε αυτό με κάποια ηρεμία και γαλήνη στη συζήτηση. Κυρία Τιεν Μαρή, είπατε κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Είπατε πολλά σημαντικά, αλλά ένα συγκεκριμένα θέλω να υπογραμμίσω εγώ. Είπατε ότι οι νέες αιτήσει είναι πιο ενδιαφέρουσες από ότι τα φάρμακα τα οποία ήδη είναι εν κυκλοφορία. Αλλά ξέρουμε λίγα πράγματα για τις νέες αιτήσει. Υπάρχουν κλινικές μελέτες, μπορεί να υπάρχουν έρευνες κτλ. Αλλά για τα νέα φάρμακα δεν ξέρουμε ποτέ αρκετά πράγματα. Ελπίζουμε ότι κάτι θα μάθουμε από, τους, ε, από τη χρήση τους ασθενείς και μόνο με την καθημερινή χρήση αυτών των φαρμάκων καταλαβαίνουμε τι καπνοφουμάρουν αυτά τα φάρμακα. Γι' αυτό χρειάζεται να υπήρχε ήδη από πάρα πολύ καιρό μια εύρωστη νομοθεσία για την φαρμακοεπαγρύπνηση, αλλά αυτή η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι χρήσιμη αν χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο κάθε ασθενής, ο κάθε ιατρός ο οποίος συνταγογραφεί ένα φάρμακο θα αναφέρει τις παρενέργειες. Και δεν ξέρει η ΕΜΕΑ αν πράγματι συλλέγει όλες τις πληροφορίες από τους <clears throat> ιατρούς. Πάντα γίνεται αυτό με ένα αποσπασματικό τρόπο και βασίζεται πολλές φορές στην τύχη. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε το τι γίνεται με τα φάρμακα και ποιες είναι οι συνέπειές τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο της ε, ε, υπηρεσίας φαρμακών. Ο Πανιόλ είπε ότι θα έπρεπε να υπάρξει περισσότερη επαγρύπνηση μέσα στα κράτη-μέλη και η κυρία Ριβάση είπε ότι δεν έκανε τίποτα η ΕΜΕΑ. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ του φορέα αυτού αν έχει πραγματικά το ρόλο που θέλουν να τους αποδώσουν ορισμένοι. Υπάρχουν αποκεντρωμένοι φορεί που δεν μπορούν να πράξουν τίποτα ω αρχέ. Θα πρέπει να πληροφορήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία μπορεί να αναλάβει δράση, να ανακοινώσει κάτι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπε και η κυρία Ριβάση, μονάχα μπορούν να δώσουν πληροφορίε η ΕΜΕΑ στην, ε, στην Επιτροπή και μετά είναι ο αρμόδιο επίτροπο, ο οποίο αναλαμβάνει. Θα πρέπει να κάνουμε σαφέ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ανεξαρτησία πραγματική σε ένα φορέα και όχι μόνο ανεξαρτησία σε εισαγωγικά σε ένα φορέα ο οποίος πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις. Τι μπορούμε να αλλάξουμε εδώ. Είπαν ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές και επαχθείς οι διαδικασίες. Και η κυρία Παρβάνοβα είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν και συγκρούσεις πολλές φορές με τις εθνικές αρχές εξακολουθούν να υπάρχουν και πάντα υπάρχουν προβλήματα γιατί όλοι θέλουν να γίνεται η έγκριση κάθε φαρμάκου σε εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό σας ρωτώ ότι μπορούμε να έχουμε 27 εθνικά συστήματα και αυτό είναι ένα καλύτερο πλαίσιο από το να έχουμε ένα μοναχά ευρωπαϊκό σύστημα. Θέλετε να διατηρήσετε 27 εθνικά συστήματα γιατί νομίζετε ότι είναι πιο εύκολο να τα ελέγχετε πιο διάφανα ή πιο ασφαλή. Αν είναι έτσι, ευχαριστώ πολύ. Με τις υγεία σας. Τότε δεν χρειάζεται να σκεφτούμε τίποτα περισσότερο αν έχετε μια τέτοια άποψη. Όλα αυτά τα οποία είναι στα εθνικά κράτη είναι πραγματικά αδιαφανή. Και βλέπετε και τους εμπειρογνώμονες στα κράτη-μέλη. Οι επιρρογνώμε θα έπρεπε σε όλε τι περιπτώσει να δηλώνουν ποια είναι τα συμφέροντά του και αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και για του πίνακε συσχετισμών, ναι, αυτή είναι χρήσιμη. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μα απασχολεί. Δεν λέμε ότι τα κράτη-μέλη ότι τα κράτη-μέλη ουσιαστικά αναλαμβάνουν για δικό του λογαριασμό την χρήση της νομοθεσίας. Τα κράτη-μέλη δεν είναι αυτά τα οποία νομοθετούν σε αυτό το τομέα, εφαρμόζουν την νομοθεσία και θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος αυτής της εφαρμογής. Πάντα έχουμε προβλήματα για να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορείτε στα χαρτιά να το προβλέψετε ότι θα γίνει κάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει στην πράξη. Αυτά είναι λοιπόν τα σημεία για τα οποία εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω ενοιολογικά προβλήματα να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο ζητούν ορισμένοι. Πάντα θα έχουμε προβλήματα με τα φάρμακα, δεν έχω καμία ψευδέστηση. Η μόνη βελτίωση, το μόνο πλεονέκτημα το μόνο ε, πλεονέκτημα το οποίο μπορούμε να αποκομίσουμε είναι ότι αν υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει ένα σημείο αναφοράς που μπορεί να ελέγχει σε όλη την Ευρώπη τι γίνεται. Και δεν μπορεί να και δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό μέσα από τις εθνικές αρχές, η οποία η κάθε μία με αυθαίρετο τρόπο η μία εγκρίνει ένα φάρμακο, η άλλη δεν εγκρίνει κανένα φάρμακο. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να προβλέψω μια τροποποίηση του καταστατικού αυτού του φορέα φαρμάκων. Εμείς θέλουμε σε όλους τους φορείς να υπάρχει κάποιος στο διοικητικό ε, συμβούλιο τους, κάποιος ο οποίος έχει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό ισχύει και για την, τροφιμική, για την υπηρεσία τροφιμικής ασφάλειας κτλ. Στο βαθμό όμως που αυτό δεν έχει ακόμα καθοριστεί, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι υπάρχουν στη, στα διοικητικά συμβούλια καταρχήν οι εθνικοί εκπρόσωποι και ουσιαστικά περνάει η εξουσία μέσα από τα μεγάλα κράτη. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι αυτοί που θα πρέπει πραγματικά να τους ε, κυνηγήσουμε και να τους διώξουμε δεν είναι το σύστημα, είναι τα κράτη-μέλη. Το ξέρεις αυτό Αντωνία. Το τελευταίο που θέλω εγώ είναι να αποδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τον οργανισμό φαρμάκων. Αν είχε κάνει κάτι το οποίο ήταν λαθασμένο, εντάξει. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ήδη δεν είχε τις δυνατότητες να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Το 1998 δεν έπαξε κάτι το οποίο ήταν λαθασμένο. Και το να συζητάμε εθνικές περιπτώσεις όπως είναι αυτή η γαλλική περίπτωση του Mediator δεν είναι λάθο να το συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί καταδεικνύει ότι πραγματικά η εφαρμογή ορισμένων οδηγιών γίνεται με λαθασμένο τρόπο. Ευχαριστώ. Η Ελίνα Μαγκάουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που ακούσαμε το ιστορικό για το Mediator πραγματικά είναι ανησυχητικά και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κενά εγώ είμαι εισηγήτρια για την ε, πιο πρόσφατη ε, νομοθεσία περί φάρμακο έτσι νιώθω κάπως υπεύθυνη. Και όταν έμαθα για το Μεντιατόρ τον Ιανουάριο, ήρθα σε επαφή με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και μου είπαν ε, ότι η νέα νομοθεσία κλείνει όλα αυτά τα παραθυράκια και όλα αυτά τα κενά. Έχουμε όμως τώρα τις δοκιμές αντοχής της Κομισιόν. Πολύ καλό το μέτρο αυτό. Και ακούμε τελικά ότι φαίνεται ότι υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν παρόλα αυτά στην νομοθεσία. Θέλω λοιπόν πραγματικά η Κομισιόν ε, να προβεί στις αλλαγές αυτές το συντομότερο δυνατό. Προτού πρέπει να εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία. Είμαστε εδώ πολλοί από τους σκιώδεις για τη νέα νομοθεσία. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Γιατί σκεφτείτε ότι αν πρέπει... Ε, έχουμε, το άρθρα εδώ, έχω μπροστά μου τα άρθρα για τα οποία μιλάμε. Και έχω δει και τα αποτελέσματα του, της δοκιμής αντοχής. Τι βρήκε ακριβώς η Κομισιόν, θα θέλαμε και εμείς να το γνωρίζουμε. Μας είπαν ενισχύουμε την νομοθεσία σε κάθε επίπεδο. Αυτό το θέλαμε και εμείς. Η Κομισιόν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων Μα έλεγαν ότι με κάθε μέτρο ενισχυόταν αυτό το σύστημα. Αν υπάρχουν θέματα ακόμα όμως, κάποια νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα, αν διαβάσω και το κείμενο που έχω μπροστά μου. Αν υπάρχει εθνική απόσυρση, να γίνει αυτόματο. Με μια-δυο μικρές αλλαγές στο κείμενο. Το ίδιο και με τη φαρμακοβιομηχανία, με τι εταιρείε. Αυτόματη απόσυρση. Νομίζω ότι θα έχουμε τις εξελίξεις αυτές πριν πούμε το ναι όλοι εδώ από όλες τις πλευρές. Να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Υπάρχουν βελτιώσεις βέβαια. Άκουσα αυτά που είπε η κυρία Παρβάνοβα για τη δήλωση συμφερόντων. Οι εθνικές διεκτυακές πύλες πρέπει να αναφέρουν κάποια, κάποια στοιχεία. Παραδείγματος χάρη δήλωση με το οικονομικό συμφερόντων, έμεσων συμφερόντων πριν από κάθε συνάντηση και αν υπάρχει ε, σύγκρουση συμφερόντων. Άρα υπάρχει βελτίωση με την νέα νομοθεσία για το θέμα της διαφάνειας και για τη σύγκρουση συμφερόντων. Και σε ό,τι αφορά τις μελέτες ασφάλειας μετά την έγκριση του φαρμάκου, επίσης έχουμε κάνει βελτιώσεις γιατί πρώτον, πρώτα ζητούνταν να γίνουν αυτές οι μελέτες, δεν γίνονταν. Τώρα είναι υποχρεωτικό. Απαιτείται από την νομοθεσία να γίνουν αυτές οι μελέτες. Και αν δεν γίνουν, υπάρχουν στον νομοθέτη ε, τα μέσα που θα του επιτρέψουν να στραφεί κατά των εταιριών. Επίσης, κατάλογος φαρμάκων που υπόκεινται σε έγκριση μετά την θέση αγορά. Και αυτά δημοσιεύονται στις δικτυακές πύλες. Καλό αυτό. Άρα θα έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Αλλά λέω, εάν υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα, α το κάνουμε πριν τεθεί σε εφαρμογή νέα νομοθεσία. Ο οργανισμό φαρμάκων ίσω να μου πει ότι ναι, ε, το επεξεργάζεται το θέμα αυτό. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε παραθυράκια, δεν πρέπει να αφήσουμε κενά. Να κλείσουμε όλα τα κενά, όλες τι τρύπε. Και αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να το κάνουν, α μα εξηγήσουν γιατί. Γιατί εμεί εδώ στο κοινοβούλιο είμαστε όλοι μαζί, απαιτούμε να κλείσουν τα παραθυράκια και τα κενά. Και να μα πει το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη γιατί δεν του ικανοποιεί αυτό, αν δεν του ικανοποιεί. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε πάλι στου προσκεκλημένους μα, δυστυχώ όμω δεν έχουμε και τόσο χρόνο στη διάθεσή μα Θα του παρακαλέσω λοιπόν να περιουστούν σε σύντομα σχόλια. Τρία λεπτό καθένα. Πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στο δόκτωρα Ετιέν Μαρία από τον Άγκας. Κύριε Πρόεδρε, γρήγορα, τάχιστα, μίλησατε πολύ για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και για τον Γαλλικό Οργανισμό και για τη ρύθμιση και και να σας πούμε ότι έχει άμεση ευθύνη ε, το εργαστήριο Σερβιέ για 30 χρόνια χρησιμοποίησε κάθε δυνατή μέθοδο για να κρύψει την πραγματικότητα, τη φαρμακολογική αυτού του φαρμάκου και τις ε, περίπτωση, τα καταπερίπτωση παρενέργειες, ε, το μειώσει το επίπεδο κινδύνου και συναγερμού και με διάφορους ε, εμπειρογνώμονες που υποσχόταν ε, αναλύσεις αλλά δεν έκαναν τίποτα, <laughs> χρησιμοποίησε οτιδήποτε μέσα από το χέρι του, μέσα του κανισμού για να αφεληθεί. Δεύτερο, θεωρώ ότι κάποια σημεία ουσιαστικά που οι διάφορες διοικήσεις και ε, στη Γαλλία θα έπρεπε να ασχοληθούμε αυτά. Έχουμε μια σύγκρουση συμφερόντων κτλ. Ξέρουμε τι γίνεται ανάμεσα στι εσωτερικέ έρευνε με εξωτερικού συνεργάτε. Επίση το κόστο και το κίνδυνο, το όφελο το, το κίνδυνο ανάλογα με την ε, προσθέμενη θεραπευτική αξία, τι γίνεται, τι συνήθειε και όσοι συμμετέχουν ε, που διαβουλευόμαστε με αυτό στη Γαλλία ε, βλέπουν αυτά τα ουσιαστικά σημεία και για να απαντήσω την κυρία Γκροστέτ ε, όλα αυτά θα εξεταστούν ε, σίγουρα βέβαια μέσω και της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Γκροστέτ και την κυρία Ρότ Μπέραντ για τις ε, παρεμβάσεις σας, γιατί τόνισαν ότι η ΕΜΕΑ βοηθάει να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό σύστημα για τα φάρμακα. Υπήρξε μια συζήτηση για το Μεδιάτορ η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα. Και που εδώ θέλω να τονίσω ότι η νέα νομοθεσία <clears throat> έχει ενισχύσει πραγματικά την φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ευρώπη. Αλλά όπως ξέρει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Μπορεί κανείς να προχωρήσει πολύ περισσότερο σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Εμείς θα πρέπει να δούμε πρωτού κάνουμε μια νέα ρύθμιση πώς ε, λειτουργεί η τρέχουσα ρύθμιση στην πράξη. Θα πρέπει να προστατευτούμε όλοι από την ψευδέστηση ότι με μεγαλύτερη φαρμακοεπαγρύπνηση στα 27 κράτη-μέλη θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε προβλήματα κρίσης. Κάθε άλλο. Εγώ νομίζω ότι αν κοιτάξουμε προσεκτικά τώρα τι γίνεται με όλα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται τώρα στην αγορά, αν έχουμε περισσότερες μελέτες που ζητάμε, αν έχουμε όλο και περισσότερες εκθέσεις που ζητούμε για όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν τύχει εθνικής έγκρισης, θα αυξηθούν οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα και όχι να μειωθούν. Γιατί τα προϊόντα τα οποία έχουν τεθεί στην αγορά ουσιαστικά υποστηρίζονται από μία αποδυναμωμένη φαρμακοεπαγρύπνηση σε εθνικό επίπεδο και μία αποδυναμωμένη διαδικασία εκθέσεων και ερευνών. Όταν βλέπουμε λοιπόν πώς έχουν έρθει όλα αυτά τα προϊόντα στην αγορά, είναι φανερό ότι οι επικρίσεις για τις διαδικασίες αυτές και για τα φάρμακα θα αυξηθούν. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τον συνάδελφό μου να πει ορισμένα στοιχεία για, το, για ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Παρακαλώ, αλλά σύντομα λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος να επανέλθω στα σχόλια που έγιναν για το Μπρίξ, για το οποίο η Επιτροπή μας την προηγούμενη εβδομάδα είχε μια συζήτηση σε βάθος και εξήτασε όλα τα δεδομένα από τη Φιλανδία, από την Σουηδία και κάποια δεδομένα επίσης από τη Γαλλία. Χρησιμοποίησαμε την αρχή της πρόληψης <clears throat> για να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που δίνονται στους ιατρούς και στους ασθενείς ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα αποτελέσματα αυτών των μελετών. Είχαμε όμως και κάποιες μεθοδολογικές ανησυχίες ότι το να το αναφέρουμε αυτό για να το αναφέρουμε αυτό σε προσωπικό επίπεδο σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει μια μελέτη κόστους ωφέλους ο ιατρός σε σχέση με τη χρησιμοποίηση αυτού του φαρμάκου για τα παιδιά και τους εφήβους. Έχουμε τώρα νέες μελέτες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες τον Ιούλιο. Η Επιτροπή μας λοιπόν κοίταξε όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα, χρησιμοποίησε την αρχή της πρόληψης, έχει συνιστήσει τροποποίησεις για την πληροφόρηση που περιέχει το προϊόν αυτό συσκευασία του και θα το επανέλθει στο θέμα αυτό τον Ιούλιο. Και η Κομισιόν για να κλείσει και παρακαλώ δύο λεπτά το μάξιμο. Σας ευχαριστώ. Τρία σημεία θέλω να τονίσω. Η φαρμακοεπαγρύπνηση, συγκρούσεις συμφερόντων και ευθύνη. Είναι μερικές φορές αναπόφευκτο να υπάρχουν παρενέργειες από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Γιατί αυτό το οποίο αξιολογούμε είναι σε κλινικές μελέτες. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικό του σώμα που αντιδρά με το δικό του τρόπο. Πρέπει να είμαστε απλώς πιο Θαραλέει όταν έχουμε αρνητικά μηνύματα για να παρέμβουμε εγκαίρως και να αποσύρουμε προϊόντα από την αγορά. Αυτό πρέπει να είναι φαρμακό επαγρύπνηση και θέλω να <clears throat> διαβεβαιώ στην κυρία Μακάουεν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός η νέα μας νομοθεσία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές όπως λέει ο κύριος Σπανιόλ. Λαμβάνει υπόψη μερικά στοιχεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καταρχήν δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να πληροφορήσει τις αρμόδιες αρχές για τις παρενέργειες. Διευρύνει την έννοια του τι είναι παρενέργεια. Γιατί και για το Mediator πολλές από τις παρενέργειες δεν γινόντουσαν σαφείς από τη συντακογραφία και δίνει στην ΕΜΕΑ αυτό το οποίο δεν είχε προηγουμένως. Ένα ρόλο για να μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή έγκριση και ένα ρόλο στην εθνική έγκριση και αυτός ο νέος ρόλος που θα έχει η ΕΜΕΑ και που θα βασίζεται στη βάση αυτή δεδομένων που θα είναι προσβάσιμη και στο κοινό για τα φάρμακα. Όταν υπάρχει λοιπόν κάποιο αρνητικό σημάδι θα μας υποχρεώνει αυτό να δρούμε αμέσως. Για την σύγκρουση συμφερόντων νομίζω τα πράγματα βελτιώνονται. Οι νέοι κανόνες οι οποίοι εγκρίθηκαν από την ΕΜΕΑ τον προηγούμενο Δεκέμβριο θα εξασφαλίσουν ότι υπάρχει πραγματική διαφάνεια σε σχέση με δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων για όλους τους εμπλεκομένους. Γιατί είναι πραγματικά αδύρυτο να πρέπει να βασίζεται σε εμπειρογνώμονε εξωτερικού η υπηρεσία φαρμάκων που έρχονται από τα εθνικά κράτη. Αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να ξέρουμε αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και σε συζήτηση με τον, ε, με τον ε, ε, Επίτροπό μου συζητούμε τις δηλώσεις συμφερόντων σε όλους τους φορείς για να ξέρουμε τι ακριβώς τι γίνεται. Το τρίτο σημείο είναι η ευθύνη. Και εγώ βασίζομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Ετιέν Μαρή για την ευθύνη. Θέλω να υπογραμμίσω και πάλι ότι μέχρι το 2004 η φαρμακεπαγρύπνηση ήταν η ευθύνη μονάχα των κρατών μελών. Αυτό λοιπόν, ξέρετε, που έκανε η η υπηρεσία μας όπως ξέρετε ήταν μονάχα ένας, όπως ξέρετε, διακυβερνητικός ρόλος. Ήταν μια ευθύνη που, όπως ξέρετε, δεν είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τώρα τι ακριβώς ήταν, ήταν μια από κοινού, ξέρετε, ευθύνη. Όχι μια καθαρά ευρωπαϊκή, ξέρετε, ευθύνη. Ευχαριστούμε. Κλείνουμε αυτό το σημείο της ημέρας της διάταξης και τη συνεδρία ακόμα κλείνουμε. Η επόμενη συνεδρία είναι 23-24 Μαΐου και το απόγευμα έχουμε επίσης μια συνεδρίαση μαζί με κοινοβούλια για το κλίμα και την αλλαγή του. Παρακαλώ πάρτε όλα τα χατιά σας και τα συμπράγκαλά σας γιατί αυτή η αίθουσα θα τροποποιηθεί στη διαταξή σας μέχρι τότε. Αν αφήσετε κάτι λοιπόν στο έδρανό σας μπορεί να εξαφανιστεί. Ευχαριστώ. Πού να με